Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το 7 της ημερήσιας διάταξης. Επιστημονικά θέματα σχετικά με τα τρόφιμα. Όπως γνωρίζετε, Πρόκειται για, μια τεχνικής φύσεως έκθεση. Ως πρόεδρος και εισηγητής θα ήθελα να σας προτείνω να δεχθούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροπολογίες σύμφωνα με το 51 του κανονισμού. Εφόσον συμφωνείτε όλοι, τότε μπορούμε να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Εάν υπάρχουν προβλήματα από μέρους σας παρακαλώ να τα παρουσιάσετε. Δεν φαίνεται κάποιος να έχει θέμα. Συνεπώς μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση ως έχει. Και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πριν όμως περάσουμε στις ψηφοφορίες, θέλω να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών νέους πολιτικούς από την Κροατία. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε. Α, εκεί στο βάθος. Καλώς ήρθατε. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες τώρα. Το πρώτο σημείο προς ψηφοφορία είναι η συμβιβαστική λύση του Συμβουλίου για την πρόταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και επαλήθευση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές. Τροποποίηση του κανονισμού. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η πρόταση. Λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα στην αντίρρηση την οποία θέτει ο κύριος Γκεμπράντι και ο κύριος Έκχαουτ για τα καύσιμα. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή η αντίρρηση, γίνεται δεκτή η αντίρρηση, μπράντι. Τώρα θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση στην Επιτροπή για την επισήμαση της χώρας προέλευσης στα επεξεργασμένα τρόφιμα, του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή η πρόταση. Ε, Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση για την πρόταση ψηφίσματος για την ετικετοθεσία ή επισήμανση της χώρας προέλευσης για τα κρέατα κτλ. Θα ξεκινήσω λοιπόν δίδοντας τον λόγο Uh, Πρώτα στον κύριο Λίζε και μετά θα συνεχίσουμε με τις πολιτικές ομάδες που έχουν συνυπογράψει. Yeah, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εκπροσωπώ τη συνάδελφο Ζόμερ που δυστυχώς ασθενεί. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω και ο συντονιστής ήδη του ΕΛΚ Ακόμα δεν είχαμε την ευκαιρία σε αυτή τη θητεία μετά τις εκλογές να συζητήσουμε αυτό το θέμα και την γεγονός ότι στην ομάδα μας ήσταν διαπόψεις. Αλλά το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στην προηγούμενη θητεία και σε διάφορες ε, ψηφοφορίες και οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν με τη συνάδελφο Ζόμερ που είναι αρμόδια για το παρόν ψήφισμα. Είναι πολύ επικριτική η θεώρησή μας ως προς το ψήφισμα και αυτό που τώρα ψηφίσαμε κατά πλειοψηφία το ερώτημα δεν μπορεί αυτή την ερώτηση να την ε, υιοθετήσει όπως έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Βέβαια είναι θεμητό να θέλουν να ξέρουν οι καταναλωτές ε, από πού ε, προέρχονται τα τρόφιμα που τρώνε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι αυτή τη στιγμή καταλάβει ο κόσμος ότι θα του κοστίσει περισσότερο. Ε, μειώνεται ραγδαία ο ενθουσιασμός ε, των καταναλωτών. Οπότε θα πρέπει να ελέγξουμε πάρα πολύ τι θα κάνουμε δεσμευτικό, νομικά δηλαδή. Εγώ καλωσορίζω να γράφουν οι εταιρείε από πού προέρχονται τα προϊόντα ε, και να αυξάνεται και η τιμή του προϊόντος, αλλά μετά αυτό είναι μια ελεύθερη επιλογή του καταναλωτού αν θα το αγοράσει ή όχι. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει αυτό να το αποφασίσουμε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια παντού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το επιβεβαιώσει και αυτή και μιλάει για ένα παράδοξο ότι οι καταναλωτές επιθυμούν με περισσότερη πληροφόρηση αλλά δεν είναι πρόθυμοι να βάλουν το γέρι στην τσέπη. Άρα, ε, τι δυνατότητες υπάρχουν αν οι καταναλωτές δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερο. Κάπου πρέπει να βρεθούν αλλού τα χρήματα. Μπορούμε να ε, διαπληκτιστούμε και για τα μεγέθη και για τα ποσά. Εγώ αμφισβητώ τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται. Είναι ένα κλάσμα και μόνο, λέει, ε, αλλά από την πρακτική εμπειρία εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό ειδικά γνωρίζω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για 50% μέχρι και 50% επιπλέον κόστος. Εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση όπως πάντα. Αν λέμε ότι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί περισσότερο ο καταναλωτής, πράγμα που δεν πιστεύω ότι πρέπει να πούμε, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι πρέπει να δώσουν αυτά τα λεφτά, π.χ. οι αγρότες. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τεράστιο ε, βάρος και πίεση προς στους αγρότες να, παράγουν όσο γίνεται πιο φτηνά και δεν νομίζω ότι πρέπει να αυξηθεί αυτή η πίεση. Έχουμε πολλά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τρόφιμα, ιδιαίτερα κρέα. Θυμίζω το θέμα τη αντίσταση στα αντιβιωτικά. Ε, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους 25.000 άνθρωποι διότι δεν τους πιάνουν τα αντιβιωτικά. Και ε, αυτό έχει να κάνει και με τη γεωργία και με τις πιέσεις και ε, μείωση των τιμών στην γεωργία και καλά θα κάνουμε να μην επιβαρύνουμε τους αγρότες. Και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι ειδικοί λέγουν ότι αν βάλουμε υποχρεωτική επισήμανση για όλα τα τρόφιμα. Αυτό θα οδηγήσει και σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είναι συγκριτικά μεγαλύτερη επιβάρυνση από ότι ε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις γιατί δεν έχουν πολύ περιθώριο και δεν πρέπει αυτό να το ενθαρρύνουμε. Ο Επίτροπος Πόρτς ε, είπε στη συζήτηση στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα ότι δεν υπάρχει, λέει, καμία σχέση ανάμεσα στην προέλευση του προϊόντος και την ποιότητα του προϊόντος. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε και στην Ευρώπη ολόκληρη ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Οπότε πρόκειται μόνο για μια ανάγκη ενημέρωσης, ε, μια επιθυμία του καταναλωτή που δεν θέλει όμως να την πληρώνει. Και αν θέλει να την πληρώνει μπορεί να το κάνει από σήμερα, εθελοντικά. Ε, τώρα υπάρχει και το θέμα της απάτης και το σκάνδαλο με το ήπιο κρέας. Αυτό είναι θέμα απάτης και είναι κακό παράδειγμα. Πρόκειται για ένα κρέας που είχε βαφτιστεί βόδι, αλλά ήταν άλογο. Για το βόλιο κρέας έχουμε πολύ αυστηρές, τις αυστηρότερες ρυθμίσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί, Παρ' όλα αυτά δεν απετράπει το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, άρα θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι και κυρίως αυστηρότερα πρόστιμα. Όπως λέει και έκθεση Ντελάνγκε και έκθεση Πυρίλο, που δίνουμε τώρα συνέχεια σε αυτήν με ε, επίσημους ελέγχους και επιθεωρήσεις και κρεοσκοπήσεις. Τώρα, αν μιλάμε για μεταποιημένα επεξεργασμένα προϊόντα, με το κρέας αλόγου ήταν η λαζάνια, έτσι δεν ήταν το κρέας σκέτο και κυκλοφόρησε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, πήγαινε έλα και τελικά κατέληξε σε λαζάνια. Και έγραφε πάνω ο κρέας. Και ποιον θα βοηθούσε αν έγραφε το λαζάνι πάνω ο κρέας προέλευση Ρουμανία, προέλευση Ιρλανδία. Παρ' όλα αυτά δεν θα τα βόλιο, θα ήταν άλογο έτσι κι αλλιώ. Οπότε είναι κακό παράδειγμα αυτό για να επιβάλλει επιπλέον και υποχρεωτικέ ρυθμίσει μα. Λοιπόν, η συζήτηση μόλι τώρα αρχίζει και ενδεχομένω και στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο θα χρειαστεί να κάνουμε συμβασμού γιατί διαφωνούμε, όπω σα είπα, μεταξύ μα. Τονίζω ότι στην περασμένη θητεία το συζητήσαμε επανειλημμένα και κατά πλειοψηφία η ομάδα μα συμφωνούσε με τη Ρενάτε Σόμερ εθελοντικά μπορεί κανείς πάρα πολλά πράγματα να κάνει και εγώ αυτό το καλωσορίζω ε, οι εταιρείε να γράφουν εθελοντικά αλλά να κάνεις δεσμευτική ρύθμιση για όλες τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες στα 28 κράτη-μέλη αυτό μας ε, προβληματίζει πολλούς από εμάς και δυστυχώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Μιλμόντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να το θέσω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το συζητήμα αυτό το θέμα εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια και εκπλήσωμαι από τα σχόλια του κύριου Λίζε. Βλέπω ότι διαβάζει τα λόγια της ε, κυρίας Σόμερ και όχι δεν μας λέει τα δικά του, διότι η άποψη του Κοινοβουλίου ήταν σαφής. Η άποψη του, του ε, το Κοινοβούλιο ψήφισε να υπάρχει αυτή η επισήμανση και κάθε φορά που υπάρχει τέτοια ψηφοφορία υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την επισήμανση του κρέατος για την προέλευση. Οπότε μου φαίνεται πολύ περίεργο που ο λέει το αντίθετα. Εκτός αν τον παρανόησα. Και αυτό ισχύει. Η προέλευση του, του κρέατος είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των ζώων, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για περιβαλλοντικά ζητήματα και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή ε, χαίρομαι που υπάρχει επισήμανση προέλευσης για το φρέσκο κρέας και οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν πλέον ε, από πού προέρχεται το κρέας στα μεταποιημένα προϊόντα. Σύμφωνα με έλεβα, το 90, το 90% των καταναλωτών θέλει αυτή την πληροφορία, να ενημερώνεται δηλαδή. Οπότε ε, είμαι πολύ απογοητευμένη από την ανακοίνωση της Κομισιόν που λέει ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν να βάλουν το χέρι ε, στην τσέπη. Δυστυχώ, η Κομισιόν χρησιμοποίησε στοιχεία από, την ίδια, από τον ίδιο κλάδο. Γι' αυτό και το, οι τιμέ που παρουσίασε στου ε, ερωτηθέντες ήταν πάρα πολύ υψηλές. Τα στοιχεία, για παράδειγμα, ε, από τη Γαλλία λένε ότι η επισήμανση του κρέατος στην, στην ε, σάλτσα μπολονέζ κοστίζει λιγότερο από ένα σέντ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το, το ποσό αυτά, ποσά αυτά και πάρα πολλέ εταιρείε ήδη επισημαίνουν τα κρέατά του στα μεταποιημένα προϊόντα. Οπότε και δυνατότητα υπάρχει και ούτε τόσο ακριβό θα ήταν. Και όσον αφορά τους ε, γεωργού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπατε για του γεωργού. Γιατί οι γεωργοί είναι αυτοί που έχουν ασκήσει τι μεγαλύτερε πιέσει για να υπάρχει αυτή η επισήμανση. Οπότε δεν λέτε αλήθεια όταν λέτε ότι δεν υπάρχει, ότι οι γεωργοί δεν θέλουν την επισήμανση. Δύο χρόνια μετά το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, οι καταναλωτές περιμένουν από τους νομοθέτες να κάνουν το σύστημα πιο διαφανές. Δεν, είναι απαράδεκτο που ακόμη δεν έχουμε αναλάβει δράση και νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων σε σχέση με το ψήφισμα αυτό και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη προς το ψήφισμα ακόμα και από μέλη του ΕΛΚ και φυσικά οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμά τους να ενημερώνονται. Εγώ θέλω να μάθω τι φοβάται η βιομηχανία κανονικά μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο σύστημα διαφάνειας θα πρέπει να το χαιρετίζουν. Όταν ε, εγώ αγοράζω ένα σάντουιτς με κοτόπουλο και μου λέει ότι είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ενώ είναι από την Ταϊλάνδη, αυτό δεν είναι διαφάνεια. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε στις νομοθετικές προτέσεις με το συντομότερο δυνατό. Η τελευταία πρόταση της, Κομισιόν κάπου βάλτωσε. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρόταση θα έρθει πιο γρήγορα. Και ε, να σας πω κάτι, το ίδιο πράγμα εύχονται και οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you very much. And now for the ECR. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν πορά να προσθέσω μετά από αυτά τα οποία είπε η Γκλένη. Την υποστηρίζω σε όλα. Ίσως εγώ ε, δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα στην απάτη με το ε, κρέας από άλογα γιατί αυτό επρόκειτο για μια ξεκάθαρη απάτη. Η απουσία λοιπόν της χώρας προέλευσης στην ε, ετικέτα και το παράδειγμα που ανέφερε η προλαλήσασα για τα σάντουιτς νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είχαμε αναλάβει την υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει σωστά μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων τους καταναλωτές. Ανέλαβαν λοιπόν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Και αυτό το οποίο πρότειναν τελικά ήταν, για να είμαι ευγενής, απογοητευτικό να υπενθυμίσω στα μέλη, τα οποία διαρωτώνται ακόμα για το αν θα υποστηρίξουν ή όχι την πρόταση, να κοιτάξουν στο τέλος του ψηφίσματος. Εκεί αναφέρεται ξεκάθαρα η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε σε βάθος τις μελέτες επιπτώσεων και να εξετάσουμε επίσης τις ε, συνέπειες σε επίπεδο της, ε, τροφι... της αλυσίδας διανομής όπως επίσης και του κόστους. Ε, το ψήφισμα δεν ασχολείται με αυτά. Το ψήφισμα μας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με την ουσία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιατενμάκη έχει το λόγο. Kiitoksia. Tämä on todella vaikea. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πράγματα είναι ε, η υπόθεση αρκετά περίπλοκη. Καταρχάς χαίρομαι που τελικά είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε για τη συγκεκριμένη πρόταση. Και ελπίζω να την υιοθετήσουμε. Τώρα, α, επί της ουσίας, είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να αναφερθούμε στην υπόθεση βέβαια του κόστους και πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Ε, στη Φιλανδία σαν παράδειγμα το κόστος το οποίο μπορεί να προκληθεί από τις αλλαγές είναι πολύ υψηλό. Ε, ενώ άλλες εταιρείες υποστηρίζουν το κόστος δεν ξεπερνάει το ένα σεντ ε, ε, για κάθε προϊόν. Συνεπώς δεν τίθεται ουσιαστικά το θέμα. Το θέμα είναι βέβαια να δούμε το πράγμα από πλευράς του καταναλωτή. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να έχει εμπιστοσύνη στα προϊόντα τα οποία καταναλώνει. Αυτό είναι η ουσία. σημασία έχει η άποψη του καταναλωτή. Κατανοώ βέβαια ότι ε, δεν ε, ενδιαφέρονται όλοι με τους καταναλωτές και το τι επιθυμούν οι καταναλωτές. Κάποιοι ίσως για τους δικούς τους λόγους θέλουν να το αγνοούν. Υπάρχει και το θέμα της ανταγωνιστικότητας και πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ε, θα εκθέσουν μεν τα περιεχόμενο τις ετικέτες, σε αυτές τις λεπτομέρειες, ίσως όμως και πολύ περισσότερες κάθε φορά. Πάντως η πραγματικότητα δεν είναι ικανοποιητική και πρέπει να αλλάξει. Είναι αλήθεια ότι ένα τμήμα των συστατικών θα είναι από μία χώρα, ε, μία άλλη, ε, ένα άλλο τμήμα από μία άλλη χώρα. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στον καταναλωτή την πολλαπλότητα των πηγών και να λάβουμε υπόψη μας και το κόστος. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι ε, εταιρείε επεξεργασίας τροφίμων και επεξεργασμένων τροφίμων γνωρίζουν από πού προέρχεται ε, το κρέας που χρησιμοποιούν λόγω ακριβώς των σκανδάλων γνωρίζουν ποιες είναι οι χώρες προέλευσης, μπορούν λοιπόν να ιχνηλατήσουν ε, σε εισαγωγικά το προϊόν το οποίο χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη. Πρέπει λοιπόν αυτές τις λεπτομέρειες να τις πούμε στον καταναλωτή. Ε, πρέπει ε, να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να περνούν όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχουν στον καταναλωτή. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, και όπως και μέσα στην Επιτροπή μας υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και κατά συνέπεια διαφορετικές απόψεις. Από ό,τι άκουσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντως δεν τους ενοχλεί η πρόταση. Ε, μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι κατά της πρότασης αυτής γιατί αλλάζουν πάρα πολύ συχνά προμηθευτές Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενημερώνουν σε μόνιμη βάση τους καταναλωτές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος σε ένα θέμα το οποίο είναι από τη φύση του περίπλοκο. Η ομάδα μου δεν έχει πρόβλημα, είναι ομόφωνη Έχουν γίνει ορισμένες συζητήσεις σε σχέση με το σημείο 8, το οποίο αφορά το πιθανολογούμενο κόστος. Εγώ θεωρώ ότι το σημείο 8 στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά από τη μέχρι τώρα. Τώρα, για την ανάγκη αναφορά σε μία μελέτη μόνο, δεν ξέρω γιατί. Ε, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα παραδείγματα της καθημερινότητας. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στις επιχειρήσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την προέλευση των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Και ίσως αν ληφθούν όλα αυτά υπόψη θα πρέπει να περιμένουμε και κάποιες ε, λεπτομέρειες σε σχέση με την ανάλυση κόστους ωφέλους. Ελπίζω πάντως να προχωρήσουμε και οι ετικέτες να γίνουν πιο λεπτομερείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Λίν Μπόιλαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ που βάλατε αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάθεση. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι η κρίση με το κρέας ε, αλόγου ε, αποτελούσε μια απάτη. Αυτό αποκρισταλώθηκε και στο νου πολλών ανθρώπων και κινητοποίησε και τις αλλαγές και πολλές φορές επηρέασε και την επιστοσύνη των καταναλωτών. Αλλά ε, στη χώρα μου το ζήτημα με το χοιρινό κρέας ε, ε, ήταν επίσης, προκάλεσε επίσης προβλήματα γιατί αυτό που θεωρούσαν ότι είναι με τις διοξίνες γιατί... Το 95% των καταναλωτών θέλουν την επισήμανση προέλευσης. Αυτό είναι παρόμοιο στοιχείο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν δεν μπορεί να ε, αποτρέψει το βλέμμα της από αυτήν την ε, επιθυμία. Και αυτό που βρήκαμε στην Ιρλανδία είναι ότι με τις διοξίνες και με το κρέας αλόγου τελικά ε, πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν να επισημαίνουν οι ίδιες τα τα προϊόντα τους, οι καταναλωτές στρέφονταν σε ε, ε, μικρά καταστήματα ώστε να μπορούν να, παρακολουθούν την προέλευση του κρέατος. Είναι λοιπόν σημαντικό το το Κοινοβούλιο να καλέσει την, κοινο, την Κομισιόν να μην αγνοήσει αυτή την επιθυμία των καταναλωτών και των πολιτών για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ε, προϊόντα κρέατος. Ευχαριστώ, Τέιλορ. Thank you, Chair. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από τον Απρίλιο του 2015 οι καταναλωτές θα ξέρουν αν αγοράζουν ένα φιλέτο που είναι ε, βόιο ε, ή χείριο ε, ή άλλο ζώο που έχει εκτραφεί το ζώο και που έχει σφαγεί. Αλλά αν αγοράσω ένα chicken και ας πούμε ή κάτι άλλο, μια εξεργασμένη μορφή μου που περιέχει κρέας δεν θα έχει ιδέα. Και μας το λένε και οι παραγωγοί συνεχώς ότι 90% των Ευρωπαίων ενδιαφέρονται για την προέλευση του κρέατος και αυτό είναι αξιοσημείωτο και θέλουν να έχουν στην ετικέτα αυτή την ε, πληροφόρηση. Αν είναι νοπό το κρέας, αν έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό, δεν αρκεί να λέμε ότι είναι κρέας που έχει παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουν περισσότερα. Ε, η σήμανση του βοήου κρέατος αναφέρει που γεννήθηκε το ζώο, που ε, επαχύνθηκε και που εσφάγει. Ε, αυτό πραγματικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Και για τον οποκριας λοιπόν και το επεξεργασμένο θέλουν να ξέρουν τον, τον πλήρη βίο του ε, ζώου από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο του λέτε ότι δεν θέλετε να πληρώσουν οι καταναλωτές την αύξηση κατά 50% όπως υπολογίζεται, αν είναι ε, δεσμευτική και υποχρεωτική αυτή η επισήμανση. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, ειλικρινά. 50% θα αυξηθεί δηλαδή κατά το ίμιση η τιμή, επειδή θα μπει μια ετικέτα. Πώς να το πω. Αυτό πιστεύω ότι είναι τελείως αβάσιμο και περιμένω να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πόσο μπορεί να το εξετάσει περισσότερο και να το επαληθεύσει αυτό. Το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου έδειξε πόσο ε, περίπλοκη είναι η τροφική αλυσίδα ε, και πόσες διαδρομές ακολουθούν τα προϊόντα και αυτό ε, Ήρξησε τις απαιτήσει των καταναλωτών ε, για να γνωρίζουν ε, αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πανάκια κατά της απάτης, αλλά η υποχρεωτική επισήμανση στον οποκρέας και στα εξεργασμένα θα υποχρεώνει τους παρασκευαστές να ελέγχουν περισσότερο τους προμηθευτές τους, γιατί τελικά θα λογοδοτούν. Άρα μπορεί να είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα αυτή ε, παραγωγής και βοηθάει αυτό και τους καταναλωτές και τους παραγωγούς για να σταματήσουν αυτοί οι ασυνείδητοι να ε, προχωρούν σε τέτοιες μεθόδους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κοφεύει. Είναι τεράστια η πλειοψηφία των καταναλωτών που απλώς θα τα θέλουν αυτές τις πληροφορίες. Και θα πρέπει τώρα η έκθεση να δώσει ε, συνέχεια σε αυτά, μάλλον την έκθεση να ακολουθήσει μια νομοθετική πρόταση για υποχρεωτική αναγραφή. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέτη. Ehm, Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Pedicini. Le carni utilizzate come ingredienti nei cibi Λοιπόν, εμείς υποστηρίζουμε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται με σωστό και ασφαλή τρόπο για την προέλευση των προϊόντων τα οποία καταναλώνουν. Αυτό θα διασφαλίσει ε, την ποιότητα των ε, τροφίμων και την ιχνηλασιμότητα των κρεάτων. Η πρόταση λοιπόν είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Γιατί είμαστε Ευρωπαίοι λοιπόν, γιατί ο καταναλωτής είναι ο απόλυτος άρχον και έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σωστά. Τι σημαίνει σωστή ενημέρωση, σημαίνει η χνηλασιμότητα. σημαίνει σωστή επισήμανση και αφορά αυτό και το νοπό κρέας και το ε, τροποποιημένο κρέας. Ξέρετε τα σκάνδαλα που έγιναν στη Γαλλία με την περίπτωση Σπαγκέρο το κρέας αλόγου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μαφία που παίρνει το κρέας από τη Ρουμανία, το πηγαίνει βόλτα στην Ολλανδία το πηγαίνει μετά στην Βόρεια Γαλλία και μετά το καταλήγει για επεξεργασία τελική στην Νότια Γαλλία. Λοιπόν, τι ζητάει ο καταναλωτής την προέλευση. Επίσης θέλουμε να γνωρίζουμε αν πρόκειται για γαλλικό, για ρουμάνικο, ουκρανικό ή κινέζικο κρέας. Έχει μεγάλη σημασία η επισήμανση λοιπόν σε σχέση επίσης και με την εγκύτητα παραγωγής του προϊόντος και εδώ τίθενται σε κλιματολογικό επίπεδο οι ανησυχίες μας. Έχουν σημασία λοιπόν. Βλέπετε εδώ για τα μεταποιημένα κρέατα τι γίνεται για τα λουκάνικα. Μέσα στα λουκάνικα βάζουν ό,τι να είναι. Δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα τα λουκάνικα. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να έχουμε ενημερωμένους καταναλωτές θα πρέπει να ορίσουμε και το περιεχόμενο. Μας λένε για το κόστος. Η Επιτροπή μας λέει ιστορίες για αγρίους. Πού τα βρήκατε αυτά. Πού τα βρήκατε αυτά. Αν πράγματι οι μεγάλες βιομηχανίες ε, αντιδρούν, ε, δεν το θέλουν αυτό γιατί χρησιμοποιούν ένα μείγμα, κάνουν ό,τι να είναι για να πετύχουν χαμηλές τιμές στις προμήθειές τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να είναι συνυπεύθυνη της κακής διατροφής να μας το πει. Εμείς θέλουμε ένα υψηλό επίπεδο ενημέρωσης του καταναλωτή και θέλουμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και θα είστε υπεύθυνοι αν οι Ευρωπαίοι απορρίψουν την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προστατεύσει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η ίδια η Ευρώπη μέσω της ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Θυμηθείτε στις 30 Σεπτεμβρίου στην ακρόασή του ο κύριος Ανδροκάητης, υπεύθυνο για την ασφάλεια της διατροφής, ανακοίνωσε σε όλους εδώ μπροστά μας ότι θα επανέλθει στο θέμα της επισήμανσης ε, του κρέατος που χρησιμοποιείται στα έτοιμα τρόφιμα, γιατί ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει ε, την προέλευση. Όλα τα λέει η δήλωση του Επιτρόπου. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο θέμα τεχνικό για την ε, μετάφραση. Με τη μετάφραση. Λοιπόν, μας τα είπε όλα ο Επίτροπος, ε, ο οποίος είπε από τις 30 Σεπτεμβρίου να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την προέλευση του κρέατος στα έτοιμα τρόφιμα. Και αυτό αφορά και τον κύριο Λίζε, αφορά και όλους τους άλλους. Ίσως η κυρία Σόμερ που δεν είναι πια εδώ δεν το είχε ακούσει τότε, αλλά έχει σημασία να το επισημάνουμε. Να έχουμε υπόψη μας ε, τον οδικό χάρτη τον οποίο μας δίδει ο Επίτροπος ε, για την Υγεία γιατί ξέρουμε μέχρι τώρα ότι μόνο το νοπό κρέας ανοιχνεύεται. Θα πρέπει να τεθεί ένα τέλος στα διατροφικά σκάνδαλα. Το 90% των Ευρωπαίων καταναλωτών θέλουν να υπάρξει αναφορά στην προέλευση. Η εκστρατεία που οργανώθηκε από, την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Καταναλωτών λέγεται «Από πού έρχεται το κρέας μου» και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση το ταχύτερο δυνατόν που θα δώσει εγγυήσεις για τη διαφάνεια της προμήθειας των υλικών και θα δώσει κίνητρα στους οικονομικούς παραγόντες να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους. Πρόκειται για ένα νέο μέσο έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εμπόδια στους απαταιώνες και ακριβώς αυτό ζητάει και η πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει πάρα πολύ επιφυλακτική σε σχέση με την υποχρεωτική επισήμανση λέγοντας ότι κοστίζει πολλά. Αυτό το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές ή κάποιοι από αυτούς και αυτές οι αριθμοί τους οποίους προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πραγματικά υπερβολικοί. Το σύστημα λειτουργεί για το φρέσκο κρέας και μπορεί επίσης να ισχύσει και για τα έτοιμα τρόφιμα. Ε, το σύστημα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ισχύει για τα έτοιμα τρόφιμα, είναι αποτυχία. Ε, στα πλαίσια μιας έρευνας που έκανε η οργάνωση και το κρέας αναφέρεται μόνο στο 48% των κατεψυγμένων προϊόντων, 29% των προϊόντων των κονσερβοποιημένων και 21% των προϊόντων σε ε, μπολ και σε ανοιχτά ή κλειστά σκεύη. Ε, και το 23% αυτών που είναι σε βάζα. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτε μας, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και θα πρέπει το ψήφισμα αυτό να γίνει δεκτό από μεγάλη πλειοψηφία ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάνι έχει το λόγο. Köszönöm szépen a Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό έχει πολλές πλευρές, υπάρχουν πάρα πολλές ε, απόψεις και νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούν ε, σφαιρικά οι καταναλωτές ε, στην Ευρώπη. Εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ευρώπης και αυτούς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε. Αυτό άλλωστε είναι και το καθήκον όλων μας εδώ. Υπάρχουν τεχνικά στοιχεία τα οποία μπορεί να εμπιστευτεί κανείς. Γνωρίζω ότι υπάρχουν παραγωγοί τροφίμων που πράγματι στην περίπτωσή τους ισχύει. Το, το, προϊόν τους θα έπρεπε να πολιθεί κατά 50% ακριβότερα αν έπρεπε να, ανα, να αναφέρουν την προέλευση του προϊόντος τους. Αλλά αυτό θα ε, οδηγούσε σε μια κατάσταση ε, να μην μπορούν οι παραγωγοί αυτοί πλέον να διαθέτουν στην αγορά φθηνό κρέας και ε, αν φυσικά δεν μπορούν να, να χρησιμοποιήσουν η παραγωγή αυτή αυτό το φθηνό κρέας, τότε θα αυξηθούν και οι τιμές των προϊόντων. Στην Ουγγαρία, σε μια σειρά από καταστήματα, μπορεί κανείς να αγοράσει κρέας φθηνότερο από 3 ευρώ το κιλό. Η προέλευση αυτού του κρέατος βεβαίως είναι ε, πολύ υποπτή. Με δύο λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν η προέλευση γίνει υποχρεωτική για το κρέας αυτό, τότε αυτό θα σήμαινε ότι πολλοί παραγωγοί που αυτή τη στιγμή εξαπατούν τους καταναλωτές, γιατί ε, παράγουν κακής ποιότητας προϊόντα, θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Και εκείνοι που θα παρήγαγαν ε, ποιοτικά προϊόντα θα τα πήγαιναν μια χαρά. διότι πρόκειται για προϊόντα για τα οποία η παραγωγή τους δεν χρειάζεται να ντρέπονται για αυτά. Η Ουγγαρία λοιπόν υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή γιατί αποστέλει και ένα μήνυμα στη βιομηχανία και στον κλάδο που θα πρέπει επίσης τέλος να καταλάβουν ότι δεν μπορούν απλά με, με τα λόμπι τους να ε, περνάει ε, να περνούν τακτικές ε, και συμπεριφορές άσχημες απέναντι στους καταναλωτές. Τελικά τι είναι ακριβό και τι είναι φθηνό. Όπως είπα, είμαι Ούγγρος και στα προϊόντα κρέατος έχουμε μια, έναν φόρο 27%. φόρους κατανάλωσης για, κρέατα, για, προϊό, για προϊόντα κρέατος. Οπότε ίσως αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει δεν είναι τόσο αν ένα κρέας ε, είναι ακριβό ή φθηνό, αλλά αυτή ευθυνό, αλλα αυτη υψηλή φορολογία και μάλιστα τώρα έχουν σκοπό να την ανεβάσουν ακόμα περισσότερο, 33%. Οπότε το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας με εξασφαλισμένη προέλευση που θα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Τελείωσαν οι μιλητές. Υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαθιουδάκη, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μας δώσει τις απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή σας και ακούμε τη συζήτηση αυτή. Uh, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπλήρωσε τη νομική της υποχρέωση να υποβάλει την έκθεσή της. Όπως θα θυμάστε ήταν ε, προϊόν συμβιβασμού όταν ε, συζητήσαμε ε, την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, τον αντίστοιχο κανονισμό. Υποβάλαμε την πρόταση αυτή, την έκθεσή μας που είναι μια έκθεση ε, περιγραφής της κατάστασης και περιμέναμε ότι, ε, όπως και έγινε, θα προκαλέσει συζήτηση. Άκουσα πολλές ε, παρεμβάσεις και θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Απαντώ σε διευκρινιστικέ ερωτήσεις, γιατί οι ερωτήσεις δεν ήταν πάντα ερωτήσεις, καμιά φορά ήταν και δηλώσει. Ιδιαίτερα για το κόστος και ε, πώς υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Ανάθεσαμε μια μελέτη για το θέμα αυτό και το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα της μελέτης συζητήθηκαν σε μια ομάδα ε, που λέγεται Focus Group και συμμετέχουν ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι οικονομικοί φορείς ε, και η παραγωγή και οι καταναλωτές και το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα της μελέτης και τα ευρήματα επικυρώθηκαν από αυτή την ομάδα όπου επαναλαμβάνω συμμετείχαν και παραγωγοί και καταναλωτές. Έγιναν ερωτήσεις για τη διαφορά του κόστους που αναφέρεται στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποια άλλα στοιχεία που αναφέρουν άλλες εκθέσεις, ιδιαίτερα η γαλλική έκθεση. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Υπάρχουν κάποιες πολύ ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο εκθέσεων. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κοίταξε τον αντίκτυπο στην αγορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε υπόψη τι αντίκτυπο θα είχε μια υποχρεωτική επισήμανση ε, ε, με αναγραφή της προέλευσης. Και επίσης έλαβε υπόψη στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που περιέχουν κρέας. Από το πιο απλό μέχρι το πιο περίπλοκο. Είναι ευρία η γκάμα αυτών των προϊόντων. Ενώ στη γαλλική έκθεση τι έγινε. Επικεντρώθηκαν σε προϊόντα βόηου κρέατος και ε, αφορούσε ε, η μελέτη την εθελοντική επισήμανση, όχι την υποχρεωτική. Οπότε προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Όταν θες να υπολογίσεις το κόστος ενός εθελοντικού συστήματος, διότι σημαίνει ότι όποιος δίνει αυτή την ε, πληροφόρηση είναι πρόθυμος να τη δώσει εφόσον είναι εθελοντικό και το βρίσκει και εύκολο. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αναφέρει στην έκθεσή μας και κάποια στοιχεία για το κόστος ε, που είναι ε, συνήθως λειτουργικό. Από 15 μέχρι 20% αύξηση ανάλογα με το προϊόν. Αλλά δεν είναι το κόστος του τελικού προϊόντος. Είναι το λειτουργικό κόστος. Υπάρχει και ένα κόστος ίχνηλασιμότητας που κυμαίνεται από 3 μέχρι 10%. Υπάρχει το γραφειοκρατικό κόστος για το επιπλέον ε, άχθος που είναι 8 με 12% του συνολικού κόστου παραγωγής του προϊόντος. Και επίσης υπάρχει και μια επιβάρηση των δημοσίων αρχών της τάξης του 10 με 13%. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι συγκρίσιμα τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, ούτε ε, μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι είναι έτσι κάπως ουρανοκατέβατα αυτά τα στοιχεία ή τα κατεβάσαμε από το μυαλό μας. Υπάρχει και το στοιχείο της προθυμίας των καταναλωτών. Ζητούν να έχουν ε, ένδειξη προέλευσης, ισχύει αυτό. Μέχρι 90% των καταναλωτών εδήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε μια ετικέτα που να επισημαίνει την προέλευση. Όταν όμως τους ρωτάς, θα ήσασταν πρόθυμοι να το πληρώσετε και όλο αυτό. μέχρι 10% ας πούμε περισσότερο θα δίνατε ή λιγότερο από 10% παραπάνω. Αυτό το 90% τότε γινόταν μέχρι και 60 με 80%. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της όλα αυτά τα στοιχεία. Θα σημειώσουμε ε, και τα όσα ακούσαμε εδώ στη συζήτηση και βεβαίως θα διαβιβάσουμε και το μήνυμα της συζήτησης που ήταν αρκετά σαφές και ε, δυνατό. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει για οποιαδήποτε δράση. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη φυσικά. Και σήμερα, συνεπώς, δεν είμαι σε θέση να σας δώσω κανένα προσανατολισμό. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω τώρα τις προθεσμίες. Α, η κυρία Βιλμότα έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. Ακόμα και με τους δικούς σας αριθμούς, οι οποίοι είναι λίγο αστήρικτοι, και μιας και οι οργανώσεις των πολιτών μου λέγουν ότι θέλουν να προωθηθεί αυτή η ρύθμιση, πρέπει να πω ότι ακόμα και αν το κόστος ήταν τόσο ψηλό, το 60 με 80% δέχονται αυτό το ανώτερο κόστος. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτείτε έτσι και αλλιώς σοβαρότερα. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι επιπλέον. Ίσως δεν έγινα απολύτως κατανοητός. Δεν λέμε ότι ακόμα και με τις αυξήσεις το 60 με 80% των καταναλωτών θέλουν να πληρώσουν. Το αντίθετο, εφόσον αυξάνεται το κόστος, τότε η επιθυμία των καταναλωτών χαμηλώνει και πηγαίνει στο 80%. 80% δεν θέλουν να πληρώσουν το επιπλέον κόστος. Eh, Καλώς λοιπόν. Τώρα η προθεσμία για τις τοπολογίες 17 Δεκεμβρίου, 12 με συμβαίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Ιανουαρίου του 2015 και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Φεβρουάριο του 2014. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, τα επόμενα σημεία μάλλον για τη 13 με 18 της ημερήσιας διάταξης αφορούν τις απαλλαγές. Όπως όλοι γνωρίζετε η διαδικασία απαλλαγής είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας αφού έχουν χρησιμοποιηθεί οι πιστώσεις γίνεται η επαλήθευση της ορθής χρήσης και ελέγχεται η ορθή χρήση και τότε χορηγείται η απαλλαγή προς το Ευρωπαϊκό Όργανο και τα άλλα όργανα για το έτος δημοσιονομικής αναφοράς. Αποφασίσαμε σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή εμείς να κάνουμε μια γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως επίσης και σχετικά με τις πέντε υπηρεσίες των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με αυτά τα οποία εμείς ασχολούμεθα. Επαληθεύσαμε λοιπόν το επίπεδο εφαρμογής, το ποσοστό εφαρμογής του προϋπολογισμού και θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι αντικειμενικά το επίπεδο αυτό είναι υψηλότατο και έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Αντιμετωπίσαμε επίσης και τα αρνητικά στοιχεία τα οποία σημειώθηκαν τα προηγούμενα έτη σχετικά με ορισμένες υπηρεσίες πριν μπορέσουμε τελικά να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Συνεπώς τώρα θα πρέπει να παρουσιάσουμε πολύ συνθετικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις πέντε εξωτερικές υπηρεσίες ε, που είναι στη δική μας αρμοδιότητα να παρουσιάσουμε λοιπόν τις, ε, ε, τις εκθέσεις αυτές, τις νομοδοτήσεις αυτές. Ξεκινώ με την απαλλαγή ε, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013, ε, τμήμα 3, εκτελεστικές υπηρεσίες και εξωτερικά όργανα. Εδώ το επίπεδο χρήσης, εξετάσαμε το ύψος χρήσης λοιπόν, και σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ επίσης και για το περιβάλλον το επίπεδο εφαρμογής ήταν γύρω στο 95% για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και 95,24% σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών. Σε επίπεδο λοιπόν εκτέλεσης μπορούμε να κρίνουμε τους αριθμούς αυτούς ε, ιδιαιτέρως ικανοποιητικούς, τα ποσοστά αυτά ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Να εκφράσουμε τη συνολική ικανοποίησή μας λοιπόν σχετικά με ένα πρόγραμμα το οποίο μας αφορά και αναφέρομαι στο πρόγραμμα LIFE. Για το πρόγραμμα LIFE φτάσαμε σε επίπεδο χρήσης 99,96% για τις υποχρεώσεις και 99,99 για τις πληρωμές. Συνεπώς λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως τα ποσά τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας από τις δημοσιονομικές αρχές. Και για την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ της Επιτροπής το επίπεδο εφαρμογής είναι 98,1% στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού για τις υποχρεώσεις και 98% αντίστοιχα για τις πληρωμές. Αναλύσαμε επίσης και εξετάσαμε προσεκτικά τα πιλωτικά και προπαρασκευαστικά προγράμματα. Πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις της ΣΑΝΚΟ. Είναι όλα σε πολύ προχωρημένη φάση και όλες οι πιστώσεις υποχρεώσεων έχουν πλήρως ε, χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι η πρώτη, το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα, να τα πω όλα μαζί και μετά θα πάρετε το λόγο αν τυχόν θέλετε. Η δεύτερη γνωμοδότηση αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ο οργανισμός αυτός τον εξετάσαμε και είδαμε ότι η διοικητική του δομή έχει πλέον ολοκληρωθεί. Υπάρχει ε, μία κάλυψη του οργανογράμματος σχεδόν πλήρης, 132 θέσεις σε σύνολο 138 και το 51% του ανθρώπινου δυναμικού ασχολείται επιτόπου με λειτουργικές δράσεις. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ καλύτερη από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο. Επαληθεύσαμε επίσης για την υπηρεσία περιβάλλοντος πως ε, οι αιτήσιοι λογαριασμοί της υπηρεσίας είναι θεμητή και τακτική. Πλέον δεν έχει υπάρξει δηλαδή πρόβλημα. Για την υπηρεσία περιβάλλοντος υπάρχει μια θετική λοιπόν γνωμοδότηση για την απαλλαγή. Ε, Το ίδιο ισχύει και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. <clears throat> Πέρα από την σωστή εφαρμογή λοιπόν του προϋπολογισμού προσπαθήσαμε να ελέγξουμε πως τα 4 πέμπτα των πόρων και στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν για τις λειτουργικές δράσεις. και επιβεβαιώσαμε επίσης και κάποια θέματα, ελέγξαμε κάποια θέματα τα οποία είχαν αναφανεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων απαλλαγών. Ε, είδαμε ότι κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση με συγκρούσεις συμφερόντων που είχαν αναφερθεί στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Φαρμάκων, του Οργανισμού Φαρμάκων, ξεπεράστηκαν με μια σειρά δράσεων οι οποίες ε, εφαρμόστηκαν μέσω της υπηρεσίας αυτής. Ε, λοιπόν, τα στοιχεία, τα τα οποία μας είχαν απασχολήσει τα προηγούμενα χρόνια ελέγχθηκαν εκ νέου και γι' αυτό συστήνουμε προς την ε, αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, να χορηγήσει την απαλλαγή για το 2013. Συντάξαμε επίσης μια γνωμοδότηση και για την Ευρωπαϊκή ε, ε, Υπηρεσία των Χημικών Ουσιών και εδώ έχει υπάρξει σωστή εφαρμογή ε, των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, δεν ξέρω τώρα αν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, να πω όμως ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορά τον οργανισμό χημικών προϊόντων είναι η έκθεση με τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ελέγξαμε ότι η υπηρεσία έκανε κάποιες εξωτερικές ακροάσεις για να βελτιώσει τις διαδικασίες για προμήθειες και διαγωνισμούς με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ενεστώτος έτους. Για όλες λοιπόν αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες και για τον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ε, νομίζω ότι διαπιστώσαμε τη συμμόρφωση με τα αιτήματα του ελεγκτικού συνεδρίου για την σωστή χρήση των πόρων που ήταν στη διάθεση των υπηρεσιών αυτών για το 2013. Συντάξαμε επίσης και ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. ελέγξαμε ότι το 74% του ανθρώπινου δυναμικού ασχολείται με επιστημονικές δραστηριότητες, συλλογή προϊόντων, στοιχείων, στατιστικών, αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος δηλαδή. Ε, διαπιστώσαμε επίσης ε, και την αύξηση των προσπαθειών της διοίκησης για διορθωτικά μέτρα ε, σε σχέση με τις παρατηρήσεις τις οποίες είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή διαδικασίες αυτοαξιολόγησης εσωτερικές μορφές αξιολόγησης και εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την ΕΦΣΑ, να συνεχίσει τον δρόμο της διαφάνειας ελέγχοντας τους τρόπους βελτίωσης ε, σε τομείς όπως ε, η ανεξαρτησία των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων όπως επίσης και το θέμα της ε, ε, προσβασιμότητας των αποφάσεων. Ε, η τελευταία γνωμοδότηση αφορά την χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Πέρα από τα στοιχεία τα σχετικά με τα δημοσιονομικά, Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είπαμε και για τα προηγούμενα, επαληθεύσαμε τις προσπάθειες τις οποίες έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης για να διορθωθούν οι προηγούμενες παρατηρήσεις οι οποίες είχαν διατυπωθεί από το ελεγκτικό συνέδριο αναφορικά με την ex post ε, επαλήθευση της ορθότητας της χρήσης των δάπανών όπως επίσης και της ε, οικονομίας ενέργειας και ενδυνάμεων στον τομέα της επεξεργασίας νέων εκθέσεων. Λοιπόν, αυτές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της δικής μας περιοχής αρμοδιότητας, αυτές αφορούν την δική μας γνωμοδότηση, συνολικά εκφραζόμεστα θετικά και ζητάμε από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή να προχωρήσει στην απαλλαγή, την χορήγηση απαλλαγής. Έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο, θα ξεκινήσω με την πρώτη συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ και τους εισηγητές και τον, και τον εισηγητή μας τον κύριο Λαβία που μας παρουσίασε την κατάσταση πάρα πολύ παραστατικά. Δεν θέλω να μπω στα στοιχεία ε, στις λεπτομέρειες, απλώς να συμπληρώσω κάπως τα όσα μας είπε ο εισηγητής μας. Και θα προσπαθήσω να κρατήσω την ίδια σειρά για, για όσους έχουν μπροστά τους τα έγγραφα, ίσως είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα γενικά για το <clears throat> ε, μεμονωμένο σχέδιο. Να πούμε από την αρχή ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του προϋπολογισμού, την εκτέλεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην υγεία και στο περιβάλλον. Ε, περίπου 100% είναι υλοποίηση και στις πληρωμές και στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Μια επικριτική ίσως παρατήρηση. Ε, διαπιστώθηκε ότι μόλις μισό της εκατό, και το τονίζω, 0,5% ε, του προπολογισμού για το περιβάλλον, το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων δαπανάτε. Από όλο τον προπολογισμό δηλαδή είναι μόνο μισό της εκατό αυτό. Και στο διορθωτικό προπολογισμό για τον ε, περσινό ε, χρόνο ήταν μόλις 0,8%. Και αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη και καθόλου δεν θα πρέπει να την καλωσορίσουμε, αλλά να εκφράσουμε τη θλίψη μας. Για τόσο σημαντικούς τομείς είναι τόσο λίγα τα χρήματα. Επίσης, συμφωνώ με τον εισηγητή. Έχω μια μικρή κριτική, μια ερώτηση γενικά προς το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί η δημόσια υγεία, ασφάλεια τροφίμων, περιβάλλον και κλίμα δεν έχουν συμπληρωθεί από κανένα σχόλιο. Γιατί είναι όλα εντάξει και βαίνουν καλώς και δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ε, ας πούμε τα θετικά τότε, να τα τονίσουμε και να τα εξάρουμε. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είμαι και μέλος, ξέρετε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εργάζομαι πάρα πολύ καλά σε αγαστή συνεργασία με τους προσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κάνουν παρατηρήσεις, συστάσεις και διαπιστώσεις που είναι πολύ χρήσιμες για τη μεταξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής, ιδιαίτερα την ενίσχυση ε, με τα κονδύλια, αλλά ακριβώς εκεί που τα πράγματα είναι καλά να τα λέμε κιόλας για τις βέλτιστες πρακτικές. Στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν με ικανοποιεί η αντιμετώπιση. Να κάνετε σχόλια και εκεί που πάνε καλά τα πράγματα, όχι όταν πηγαίνουν μόνο στραβά. Κάτι άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς είναι ότι το περιβάλλον και η δημόσια υγεία και ανάπτυξη της υπαίθρου και η αλληλεία είναι μαζί. Εκεί έχουμε ποσοστό σφάλματος 6,7% ενώ το γενικό ποσοστό συνήθως είναι 4,7% και αυτά τα σφάλματα κυρίως είναι στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αλία και σε καμία περίπτωση στην περιβαλλοντική πολιτική και στην πολιτική της δημόσιας υγείας. Και δεν θέλω να δημιουργηθεί στρεβλή εντύπωση και σφαλμένη εικόνα στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό, να πω σε σχέση με αυτό και πάλι, γιατί το ακούμε και από συναδέλφους εδώ ε, που κάνουν λάθος δηλώσεις στον τύπο και λάθος δημοσιεύματα. Το ένα ποσοστό σφάλματος δεν σημαίνει ότι είναι αξιόπινες ε, πράξεις, ξέρω εγώ, διαφθορά, απάτη κτλ. Μπορεί να είναι και σφάλματα και λάθη κανονικά. Ε, όταν αυξάνεται το ποσοστό σφάλματος δεν σημαίνει αποτυχία κατά ανάγκη. Μπορεί να σημαίνει και επιτυχία, δηλαδή ότι τα βρίσκουμε. Ότι κάνουμε καλύτερους ελέγχους και αποκαλύπτονται αυτά. Δεν σημαίνει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και ελέγχουμε εκεί που στο παρελθόν ήταν μεγάλος ο κίνδυνος φαλμάτων, άρα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι με τα κράτη-μέλη και ανακαλύπτονται και αποκαλύπτονται περισσότερα και ε, προλαμβάνονται. Για τις, τους υπόλοιπους οργανισμούς να πω, ε, έτσι προεξοφλώντας, ότι συμφωνώ με τις συστάσεις του εισηγητού μας, ε, να συστήσουμε απαλλαγή για όλους τους οργανισμούς και να τονίσω και πάλι θετικά ότι η διαδικασία ε, ε, του Κέντρου Ελέγχου και ε, Πρόληψης Νοσημάτων ήταν ο μόνος οργανισμός που απάντησε στη στάση του Κοινοβουλίου και αυτό μας χαροποιεί διότι φαίνεται ότι εκτιμούν το έργο μας και δίνουν συνέχεια. Και σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ε, μια μικρή παρατήρηση. Ο εισηγητής εδώ είπε ότι το 2013 χρειάστηκε έκτακτη ε, εισφορά για τα φάρμακα ε, κατά των σπανίων νόσων. Αυτό θα πρέπει να το χαιρετήσουμε και υπάρχει και αντίστοιχη τροπολογία δικιά μας, διότι πιστεύω ότι οι σπάνιες ασθένειες είναι κάτι το οποίο αξίζει πάντα την προσοχή μας και δεν περιτεύει καθόλου αυτή η προσπάθεια. Μια μικρή ερώτηση έχω τώρα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ΕΧΑ. Το 2013 ε, υπήρξε και πάλι ε, μία έκτακτη ε, εισφορά άπαξ των Νορβηγών για τα βιοκτώνα για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τι είναι αυτό, θα μπορούσατε λίγο να μας εξηγήσετε. Και σε σχέση με την ΕΦΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων, μου διέφυγε εμένα, όπως και άλλων συναδέλφων, ότι ε, μας είχαν επιστήσει την προσοχή για το εξή γεγονό, το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος μου. Για την ανεξαρτησία που για μας είναι ένας παράγον πάρα πολύ σημαντικός και η διαφάνεια αλλά και η ανεξαρτησία στο παρελθόν είχαν εκφραστεί κριτικές, όπως ακούσαμε από πλευρά ΕΦΣΑ. Έχει κάνει προσπάθειες ο οργανισμός να διασκεδάσει αυτές τις ε, επιφυλάξεις και να υιοθετήσει νέους κανόνες για τη διαφάνεια. Αλλά παρόλα αυτά, ακούμε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων σε μέλη του πάνελ που είναι του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή, Μπορεί, ο ενδιαφερόμενος λέει, μπορεί να συνεχίσει ε, να ασκεί τα καθήκοντά του γιατί δεν υπάρχει πάντα συμβίβαστο. Ε, μου φαίνεται κάπως επιπόλαια αυτή η εξήγηση και τσαπατσούλικη. Μπορείτε να με ενημερώσετε περισσότερο τι ισχύει και ευχαριστώ πολύ. Καλή συνεργασία είχαμε. Σταματώ εδώ. Κύριος Γερμπράντη. Yes, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε εσά προσωπικά για το γεγονός ότι αντικαταστήσατε τον ε, Utah Hawk, τη Utah Hawk που το έκανε αυτό για αιώνες αλλά πραγματικά τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Δεν θα επαναλάβω όσα είπατε εσείς, όσα είπε και η Καρν Κάντεμπαχ γιατί συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν. Δύο ζητήματα θα ήθελα να θέσω. Πρώτα απ' όλα Υπάρχει το γενικό πρόβλημα που έχουμε διαπιστώσει εδώ και πολλά χρόνια στην διαδικασία απαλλαγής και στις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ανησυχούν περισσότερο για να πάρουν τα χρήματα παρά για την ε, ποιότητα των έργων στα οποία τα χρήματα αυτά καταλήγουν. Και ένα από τους λόγου είναι το γεγονός ότι ε, εργαζόμαστε με αυτές τις εθνικές ε, κατανομές και προτού, προτού διανεμηθούν τα χρήματα έχουν ήδη κατανεμηθεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Και έχουμε διαπληκτιστεί με το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Current Life για να περιοριστούν αυτές οι εθνικές κατανομές όσο το δυνατόν περισσότερο και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο γενικά το αποκαλούν χρήση use it or lose it. Χρησιμοποιήστε το ή χάστε το. Αν κάποιο κράτος μέλος λοιπόν δεν αξιοποιήσει τα χρήματα τότε τα χάνει. Και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που ένα κράτος μέλος θέλει να του συμβεί. Είναι όπως όταν λέω στα παιδιά μου ότι μπορούν να έχουν ε, γλυκά αλλά μόνο αν τα φάνε μέσα σε μια ώρα. Θα το κάνουν ακόμα και αν ε, δεν τους αρέσει πάρα πολύ ή δεν τα θέλουν τόσα πολλά, θα το κάνουν μέσα σε μια ώρα. Και αυτό κάνουν και τα κράτη-μέλη. Το κάνουν για να δαπανίσουν τα χρήματα και όχι για την ποιότητα των έργων. Και παρότι στον τομέα του περιβάλλοντος αυτό, αυτές οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες, εξακολουθούν να υπάρχουν και ε, θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά με τη βοήθεια σε τελική ανάλυση και των ίδιων των κρατών μελών. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν αφορά μόνο την ετήσια έκθεση του ελληνικού συνεδρίου και αυτή τη διαδικασία απαλλαγής, αλλά Μιλώ και για την ειδική έκθεση για την βιοπικιλότητα που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το ελεγκτικό συνέδριο γιατί ε, είναι επικριτική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε τα χρήματα για τη βιοπικιλότητα. Η αποτελεσματικότητα των έργων δηλαδή που χρηματοδοτούνται δεν ε, είναι πάντοτε δεδομένη. Και το πιο ε, έντονο σημείο κριτικής είναι ότι δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς χρήματα δαπανούμε για την βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ποιο είναι τα χρήματα του προϋπολογισμού που καταλήγουν σε αυτό το σκοπό και δεν έχουμε ιδέα για το τι, τι, κονδύλια και τι χρήματα δαπανώνται στα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ε, ότι χρειαζόμαστε περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ε, κατ' έτος, ε, στο Natura για να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει, αλλά δεν έχουμε ιδέα για το τι γίνεται. Το ερώτημά μου προς την Επιτροπή είναι το εξή. Δεν είναι δική σας ευθύνη όταν θεσπίζονται κάποιοι στόχοι και σε αυτούς ε, αποδίδονται και κάποια χρήματα του προϋπολογισμού να γνωρίζουμε ποιος ακριβώς είναι ο προϋπολογισμός, ποια είναι τα κονδύλια τόσο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και στους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς. Μέχρι σήμερα ε, ελπίζουμε ότι λόγω της ε, σύμβασης για την βιοποικιλότητα που συνήθισε στην Νότια Κορέα τον προηγούμενο μήνα, όπου όλα τα συμβαλόμενα μέρη ήταν υποχρεωμένα να υποβάλουν δικές τους εκθέσεις ότι στο τέλος θα καταφέραμε να περάσουμε από την διαδικασία του ΟΗΕ και να ε, καταλήξουμε στο ποια είναι τα ποσά τελικά που δαπανώνται στα κράτη-μέλη μας αλλά ούτε εκεί τελικά καταφέραμε να μάθουμε πόσα χρήματα τελικά δια, δαπανώνται. Οπότε το ερώτημα προς την Κομισιόν είναι το εξής. Μπορείτε να μας διαθέσετε τα στοιχεία, μπορείτε να αναγκάσετε τα κράτη-μέλη να δημοσιοποιήσουν πόσα χρήματα δαπανούν για τη βιοποικιλότητα. Γιατί ξέρω ότι στη χώρα μου, στις κάτω χώρες, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ε, περιοριστεί, ε, έχει περιοριστεί ο προπολογισμό για τη φύση ε, κατά περισσότερο από 60% και φοβάμαι ότι το ίδιο έχει συμβεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να γνωρίζουμε το στοιχείο αυτό, Προτού συνεχίσουμε την, ε, στη συζήτηση ε, για την απαλλαγή και τους μελλοντικού ε, προϋπολογισμούς. Οπότε αυτή είναι η έκκλησή μου προς την Κομισιόν, να αποσαφηνίσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Κονέτσινα. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί νομίζω ότι Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν το έγγραφο γνωρίζουν ότι ε, δουλέψατε πολύ σκληρά. Υπάρχουν τόσοι πίνακες, τόσα αριθμητικά στοιχεία, εκατοντάδες σελίδες, οπότε φαίνεται ότι πραγματικά πρέπει να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο η σύνταξη αυτής της έκθεσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Κοιτάζοντας τα συμπεράσματα, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για ένα θέμα. Είμαι ε, σημείο επαφή για το ECDC και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόσληψης Νοσημάτων εργάζεται πολύ σκληρά και προσπαθούν να εξασφαλίσουν και την απαραίτητη χρηματοδότηση και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες σε αυτό, διότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς επιδημίες κτλ. Οπότε πρέπει να διαχειρίζονται τα κονδύλια τους με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δεν γνωρίζουν ποια θα είναι ακριβώς η κατάσταση σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες. Το ECDC λοιπόν έχει συμπεριληφθεί σε έναν δεύτερο γύρο ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση είναι υψηλή ποιότητα. Υπάρχουν και κάποιες συστάσεις και είμαι σίγουρη ότι ε, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόσληψης Νοσημάτων θα ανταποκριθεί στις συστάσει αυτές. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το κέντρο αυτό βρίσκεται στο σωστό δρόμο, αλλά μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε και εδώ στην Επιτροπή αν αυτό το κέντρο θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο φιλόδοξο ως προς του. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι αρμοδιότητες του είναι κάπως περιορισμένες. Αν θέλουμε ε, να συνεργαστούμε και με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα, με την Ουκρανία ή τη Μολδαβία, θα πρέπει να δώσουμε στο κέντρο αυτό την απαραίτητη εντολή και θα πρέπει να εξεύρουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Αυτά τα λέω για το μέλλον. Και πάλι να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την έκθεση αυτή, γιατί εμείς τη διαβάσαμε την έκθεση αυτή, αλλά δεν ήταν ε, δική μας υποχρέωση να κάτσουμε να την συντάξουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφο Σέβη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υπάρχει ένα επιχείρημα πάντα που λέει ότι ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, έχουμε κάποια θέματα και όταν πρόκειται για χρήματα ε, δεν μας πολύ απασχολούν. Μας απασχολούν όμως διότι είναι χρήματα των φορολογουμένων. Εγώ θέλω να μιλήσω για την ασφάλεια τροφίμων, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΕΦΣΑ. Σας είπα ε, και προηγουμένως ότι είναι χρήματα των φορολογουμένων. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί επειδή ε, πληρώνουν ε, αυτά τα χρήματα οι φορολογούμενοι. Οι δαπάνες πώς είναι εκεί στους οργανισμούς, θα πρέπει να λογοδοτούν. Γενικά συμφωνούμε με τη γνωμοδότησή σας, έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά, αλλά ε, ίσως θα μπορούσε ε, κάτι να διορθωθεί. 61 εκατομμύρια είναι 0,52 ε, ε, του συνολικού προϋπολογισμού, αλλά ε, πρέπει να έχουμε ποιοτικά στοιχεία για να ενημερώνουμε τους πολίτες. Είναι σημαντικό να ενημερώνει σωστά, δεν είναι τυχαίο. Και για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Τροφίμων, πώς καταρτίζονται οι ομάδες εργασίας. Είναι όλα αυτοί πραγματικά ανεξάρτητοι γιατί ακούγονται πολλές επικρίσεις. Είναι αβάσιμες αυτές, είναι δικαιολογημένες, τι γίνεται. Υπήρξε και ομάδα εργασίας που ήταν αρμόδια για να μετράει την τοξικότητα κάποιων ουσιών στα τρόφιμα και ανατέθηκε σε κάποιον που στο παρελθόν δούλευε στην Pepsi Cola και στη Φίλιπ Μόρις. Ε, αυτά λοιπόν θα πρέπει να ελέγχονται οι τοξικολογικές ε, εργασίες και εξετάσεις από τέτοιους ανθρώπους. 80 εκατομμύρια ήταν ας πούμε μια δαπάνη εκεί ε, και τελικά πληρώθηκε ένας εμπειρογνώμονας που ήταν στο παρελθόν υπάλληλο της Φίλιπ Μόρις και τον πήραμε στην Εύσα και κάνει μελέτες. Η σύγκρουση συμφερόντων είναι αυτή. Τελικά όπως και έλεγε το ψήφισμα του προηγούμενου Απριλίου, εμείς θέλουμε η υπηρεσία να κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα ανεξαρτησίας, δεκτικότητας, σωστής χρήσης των ποσών τα οποία έχει στη διάθεσή της. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Θα δώσω το λόγο πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος θα δώσει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τους συναδέλφους. Κάποιες από τις ερωτήσεις τέθηκαν στην ΕΦΣΑ. Αργότερα θα έχουμε μια πιο διαρθρωμένη συζήτηση με τον Διευθυντή της ΕΦΣΑ. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή είναι και την παρουσίαση σαφέστατη και ε, πάρα πολύ ακριβής για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που έγιναν. Πρώτον, για το κλίμα και το περιβάλλον, γιατί αυτές τις δύο γενικές διευθύνσεις εκπροσωπώ. Είναι γεγονός ότι είναι χαμηλό το ποσοστό του κοινοτικού προπολογισμού που αφιερώνεται εκεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα κονδύλια, υπάρχουν και άλλα κονδύλια για το περιβάλλον και για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, την έρευνα, τα διαστατικά ταμεία κτλ. Οπότε, και το είπε και ο κύριος Γκερμπράντι αυτό, αποφασίσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακολουθούμε καλύτερα το σύνολο αυτό των δαπανών στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να ε, θεσπίσουμε ένα σύστημα ίχνηλασιμότητας ε, των δαπανών και στην κλιματική αλλαγή, κυρίως ε, από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και στη βιοπικιλότητα. Αυτό ήδη θα μας επιτρέψει ε, να ε, κάνουμε τις εκτιμήσεις μας, γιατί είναι αρκετά δύσκολο αυτό μεθοδολογικά. Δηλαδή ένα έργο πώς ευνοεί τη βιοπικιλότητα, ε, πλήρως, εν μέρη, καθόλου κτλ. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Για να δίνει στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2015, γιατί το 2014 άρχισε να τρέχει νέα προγραμματική περίοδος και θα παρουσιάσουμε μια μεθοδολογία που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Επίσης, αναφερθήκατε στην ειδική έκθεση για τη βιοπικιλότητα, η οποία μόλις δημοσιεύτηκε και θα είναι και αντικείμενο συζήτησης και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και ε, σε σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου που πηγαίνει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση να προσπαθήσουμε να ε, καθορίσουμε ποια χρήματα πηγαίνουν στην βιοπικιλότητα. Ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε ήταν οι εθνικές ε, κατανομές. Το ελεγκτικό συνέδριο το επέκρινε αυτό, όχι στην έκθεση για την απαλλαγή, αλλά για την ειδική έκθεση για το πρόγραμμα LIFE και περιβάλλον. Δεν γινόταν καλή επιλογή των έργων στην κατανομή στα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί αυτό το σύστημα από το 2014 για το νέο πρόγραμμα LIFE και καταλήξαμε σε μια σταδιακή ε, εγκατάλειψη του συστήματος για να βελτιωθεί η ποιότητα των έργων. Να πω επίσης ε, κάτι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε την πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού ετήσεων στο live. Ήμασταν στα 600 με 700 όταν άρχισε το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το 2015 ε, μόλις έκλεισε ο διαγωνισμός και λάβαμε πάνω από 1300 έργα. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα επιλογής. Φυσικά δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα γύρω στα 200 ετησίως, άρα θα πρέπει να γίνει μια επιλογή εκεί αρκετά σημαντική. τα ε, θέματα που είχα να σας πω για το περιβάλλον και το κλίμα πάνω κάτω είναι αυτά. Αυτά είχα σημειώσει. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κάποιος άλλος εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Ε, από την DG Sanko, Γιώργη Λατενζημένο. Νομίζω ότι τα σχόλια που έγιναν για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων θα ήθελα να αναφέρω ότι η έκθεση του εισηγητή είναι πάρα πολύ σαφής για, αυτά τα δύο, για αυτούς τους δύο τομείς. Κατά τη γνώμη μου δεν, έχουν, δεν περιέχουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τα έργα, για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τον οργανισμό που, ε, που τους οργανισμούς ε, που παρακολουθεί η DG Sanko, η EFSA, η CDC, η EMA. Ξέρω ότι θα υπάρξει και ακρόαση με τον, ε, όσον αφορά την ΕΦΣΑ με τον κύριο Ουρλ, οπότε θα μπορείτε, αν, υπάρχει, αν υπάρχουν ερωτήσεις, να τις συζητήσετε μαζί του ε, στο επόμενο θέμα. Αυτά από μένα, ευχαριστώ. Εντάξει. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να περάσουμε στο επόμενο σημείο προβλέπει η μερίσια διάταξη μια προθεσμία για τις τροπολογίες 11 Δεκεμβρίου. 12η μεσημβρινή προβλέπεται στις 29 Ιανουαρίου η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού στις 23 και 24 Μαρτίου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε όπως είπα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, Εξάμεινο Συντονισμού. Θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και γύρω από την πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Γραμματικάκης. Δίδω το λόγο λοιπόν στον κύριο Γραμματικάκη για να μας παρουσιάσει τις θέσεις του. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου ε, γιατί έχω εντυπωσιαστεί από μέχρι τώρα δουλειά των Επιτροπών και αισθάνομαι ένα δέος για τη δική μου γνωμοδότηση. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να ανταποκριθώ σωστά γιατί είναι γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ξεκινά κάθε φθινόπωρο με την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη είναι αυτό ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής ε, των κρατών μελών, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γεννήθηκε βέβαια μέσα στην κρίση και είναι ένα από τα διδάγματα της κρίσεως. Κατανοήσαμε δηλαδή ότι αν θέλουμε η Ένωση να επιβιώσει αλλά και να δυναμώσει, αυτό θα γίνει μόνο μέσω βαθύτερης συνεργασίας και συντονισμού. Είναι πάντως αλήθεια ότι ως Ένωση έχουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες. Σχεδόν όμως αποκλειστικά θα συμφωνήσετε στη δημοσιονομική πειθαρχία και τους μακροοικονομικούς δείχτες. Αυτά όμως δεν είναι αρκετά για την αναζωογόνηση της οικονομίας, την καταπολέμηση της ύφεσης και κυρίως, το υπογραμμίζω, για την ενσωμάτωση στην κανονική ζωή των εκατομμυρίων ανέργων. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι άνεργοι αυτοί αποτελούν ήδη το 21ο κράτος της Ένωσης και πρέπει να ενσωματωθούν. Δεν είναι λοιπόν περίεργο, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι ευρωσκεπτικιστές, έστω και άδικα, κερδίζουν διαρκώς έδαφος και οι πολίτες της Ευρώπης διαδηλώνουν ακόμα και εδώ, στις Βρυξέλλες, δηλαδή στο θεσμικό κέντρο της Ευρώπης. Είναι λοιπόν φανερό ότι λείπει μια πραγματική κοινή στρατηγική για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε αυστηρούς κανόνες στα δημοσιονομικά με ελέγχους και κυρώσεις, αλλά μόνο χαλαρό και φοβούμε εν μέρει εθελοντικό συντονισμό των στόχων της στρατηγικής 2020 όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας. Ειδικότερα οι στόχοι της Επιτροπής μας που εστιάζουν βέβαια στην προστασία του περιβάλλοντος και κάνουν σπουδαίο έργο, αλλά και την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση πόρων, συχνά έχω την αίσθηση ότι παραμερίζονται, ενώ είναι αυτοί που θα βελτίωναν ουσιαστικά την καθημερινότητα του πολίτη και τις προοπτικές του για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημοσίας Υγείας ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής να θέτει στο ίδιο επίπεδο τη δημοσιονομική πειθαρχία με τη στρατηγική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρώ δηλαδή ότι η Επιτροπή μας πρέπει να έχει ένα από τους πρώτους λόγους. Διότι μόνο το όραμα ενός μοντέλου βιώσιμης οικονομίας και όχι η μείωση του κόστου εργασίας όπως ισχυρίζονται κάποιοι και ήδη διαψεύδονται μπορεί να αποδώσει στην Ευρώπη τη χαμένη ανταγωνιστικότητά της αλλά και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και πλούτο στα σύνορά μας. Επιπρόσθετα, να προστατεύσει το περιβάλλον και να προσφέρει στους πολίτες μια ποιοτικότερη, δηλαδή καλύτερη ζωή. Συνοπτικά, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει για φέτος τρεις στόχους στην ετήσια επισκόπηση – Πρώτον, τη συντονισμένη προώθηση των επενδύσεων. Δεύτερον, την ανανέωση της δέσμευσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Και τρίτο, τη λεγόμενη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Η διαφορά βέβαια με τις προηγούμενες επισκοπήσεις είναι βέβαια το πρώτο σημείο που αφορά την προώθηση των επενδύσεων μέσω του, τα έλεγα, ικανοποιητικού χρηματοδοτικού πακέτου που ήδη παρουσιάστηκε. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για μας, το Ευρωκοινοβούλιο, να απαιτήσουμε οι γενικές προτεραιότητες του επενδυτικού πακέτου να διαμορφωθούν και με τη δική μας συμβολή. Πρέπει να επιμείνουμε ότι το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής θα πρέπει να εξυπηρετεί μια στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, το υπογραμμίζω, η οποία θα ενταχθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, με συγκεκριμένους βέβαια στόχους αλλά και δείκτες ακόμα στη δέσμευση της Επιτροπής για νομοθετικές πρωτοβουλίες όπου θα χρειαστούν, όπως για παράδειγμα στο νέο πακέτο για την κυκλική οικονομία. Είναι σαφές ότι χωρίς πιο ισχυρές επενδύσεις σήμερα θα είναι αδύνατο να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και επίσης τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους του 2030 έτσι φοβούμαι ότι η Ευρώπη θα κρατηθεί κάτω από το αναπτυξιακό δυναμικό της και θα στερήσει από μια ολόκληρη γενιά τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί στη βάση της καινοτομίας και της γνώσης και όχι όπως σήμερα σε μεγάλο βαθμό του εργατικού κόστους. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλοί και ισχυροί λόγοι γιατί πρέπει η βιώσιμη οικονομία να έχει προτεραιότητα. Θα αναφέρω ενδεικτικά και με συντομία του χρόνου μόνο μερικούς. Πρώτο, κάθε χρόνο ξοδεύονται πάνω από 500 δις ευρώ για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι πόροι χρηματοδοτούν όμως κράτη με αντικρουόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα, καμιά φορά και δραματικά αντικρουόμενα ενώ θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τις επενδύσεις βέβαια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που και ποιοτικέ θέσεις εργασίας δημιουργούν αλλά και εξαγωγικό δυναμικό. Δεύτερη ενδεικτική παρατήρηση. Σε μια παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία όπως ζούμε σήμερα τα αναπτυσσόμενα κράτη δημιουργούν πιέσεις στη ζήτηση σημαντικών πρώτων υλών ανεβάζουν έτσι την τιμή τους και ασκούν αφόρητες πιέσεις σε ένα ήδη εύθραστο περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε την οικονομία μας σε ένα κυκλικό μοντέλο, όπου σχεδόν τίποτα δεν θα πηγαίνει χαμένο και εννοείται ότι το όφελος τότε θα είναι τεράστιο. Κάποιοι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι βελτιώση στην αποδοτική χρήση των πόρων θα μπορούσαν να μειώσουν τις ανάγκες ισρών υλικών κατά 17 έως 24% ένα μεγάλο ποσοστό μέχρι το 2030. Παράλληλα, η καλύτερη χρήση των πόρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολικό δυναμικό εξοικονόμησης ύψους ίσως και 630 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ευρωπαϊκή βέβαια βιομηχανία. Τρίτο, αν θέλουμε, που νομίζω ότι πρέπει να θέλουμε, να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής οικονομίας, είναι ανάγκη να πάυσουμε να πιέζουμε το εργατικό κόστος όπως δυστυχώς μέχρι σήμερα. Αντίθετα θα πρέπει να γίνουμε πιο αποδοτικοί ενεργειακά, να χρησιμοποιούμε δηλαδή πιο έξυπνα τους πολύτιμους πόρους. Τελειώντας κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ να μου επιτρέψετε για λίγο αλλά με έμφαση στη φορολογική πολιτική θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί έναν απόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και ένα βασικό εργαλείο κινήτρων και αντικινήτρων στην οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε σε φόρους που επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικά βλαβερές ενέργειες και δραστηριότητες και να περιορίσουμε αισθητά την μεγάλη έως ε, σήμερα φορολόγηση της εργασίας. Η πολιτική αυτή απαιτεί ασφαλώς ένα σύνολο, τολμηρό σύνολο μέτρων αλλά και ρήξης. Είναι όμως απαραίτητη αν πρόκειται το οικονομικό μας μοντέλο να αποκτήσει καλύτερες προοπτικές. Είναι χαρακτηριστικό, το γνωρίζετε, ότι η πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας που είναι νομίζω σωστή στις γενικές γραμμές της έχει αδρανοποιηθεί στο Συμβούλιο λόγω του κανόνα του υπάρχοντος της ομοφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση νομίζω για τη διαμόρφωση μιας κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης που θα στηριζόταν σε μια στενότερη συνεργασία όσων τουλάχιστον είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού μοντέλου. Είναι ευνόητο κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάλφοι ότι η σημερινή μου γνωμοδότηση πρέπει και το τονίζω αυτό να εμπλουτιστεί με τις δικές σας πολύτιμες ιδέες και προτάσεις ώστε η τελική μορφή της να αποτελεί ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο για αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πακτήσει ουσιαστικότερο περιεχόμενο αλλά και θα συνιστά, το τονίζω αυτό, και ένα ευίωνο σημείο για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ. Όχι. Όχι, όχι, δεν θέλει το λόγο η κυρία Γκέρλινγκ. Ο κύριος Φαρία. Ε, grazie, Presidente. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γραμματικάκη. Πράγματι πρόκειται για ένα θέμα περίπλοκο και είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την ανάπτυξη της οικονομίας από το 2015 και μετά. Το θέμα είναι να υπάρξει μια μορφή ανάπτυξης ανταγωνιστική, η οποία να οδηγήσει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης με μόνιμους όρους. Απαιτούνται λοιπόν προσπάθειες και στον τομέα των επενδύσεων, απαιτείται μια επένδυση σε εισαγωγικά εδώ σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει οι επενδύσεις να συγκεντρωθούν σε ευαίσθητους τομείς που θα επιτρέψουν την βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών δικτών. Θα πρέπει να επενδύσουμε επίσης και στην κατάρτιση και σε ένα σύστημα πληροφορικό ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο και έτσι ίσως να έχουμε και δυνατότητες περισσότερες από ό,τι σήμερα και στην παροχή υπηρεσιών και στις μεταφορές. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τον δεύτερο πυλώνα τώρα, τις διαρθρωτικές αλλαγές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο να είναι πιο ευνοϊκό για τις επενδύσεις μέσω σαν παράδειγμα της, ε, της κατάργησης των εμποδίων για την είσοδο στην αγορά. Απέναντι σε αρνητικές μορφές ανάπτυξης ε, χρειαζόμαστε ένα σύστημα διακανονιστικό το οποίο να σέβεται τις επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός και στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και συμφωνώ με τον εισηγητή ε, για την ανάγκη ε, ύπαρξη συστημάτων προνοίας, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, υψηλής ποιότητας και βιώσιμων οικονομικά. Είναι μια ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα άλλωστε και προσφέρει και πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης. Στον τομέα των δημοσιονομικών πολιτικών πολλά μένει να γίνουν. Οι προϋπολογισμοί πρέπει να καταστούν πιο ευνοϊκοί για την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη πάντα και την αηφορία. Θα πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί αντιστάθμισης και μέσω του σεβασμού του περιβάλλοντος, μέσω της φορολογίας πράσινου σε εισαγωγικά τύπου, απαιτείται ένα καλύτερο σύστημα ε, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων απορριμμάτων και θα πρέπει να βοηθήσουμε την βιομηχανία να βρει τρόπους ε, ε, επεξεργασίας των αποβλήτων αντισταθμίζοντας το επιπλέον κόστος όπου αυτό χρειάζεται. Πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδιαίτερα στους τομείς οι οποίοι δεν φύγουν άμεσα τα δημοσιονομικά. Θα πρέπει να εντάξουμε και πληρέστερα τη στρατηγική 2020, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, την παινία και, την, και στηρίζοντας την αηφορία. Θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις στις απαιτούμενες σε εθνικό επίπεδο επίσης μεταρρυθμίσεις, αλλά συγκλίνοντας ε, ε, σε επίπεδο κοινοτικό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν αυτό το στόχο. Θα καταθέσουμε λοιπόν ορισμένες τροπολογίες και για μια ακόμη φορά ευχαριστώ πολύ τον κύριο εισηγητή. So... Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Κυρία Κόνιτσνα. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το γεγονός ότι ανέλαβε αυτό το έργο. Αλλά όπως είπα και το Σεπτέμβρη φέτος, όταν συζητήσαμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα για άλλη μια φορά. που θεωρώ ότι λείπουν από την έκθεση αυτή και θα ήθελα με κάποιον τρόπο να συμπεριληφθούν ως σκιώδης εισηγήτρια. Χαιρετίζω τα λόγια του συναδέλφου που είπε ότι είναι απαραίτητο να οριστικοποιηθεί η γνωμοδότηση αυτή και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σε πνεύμα συνεργασία. Το πρώτο πράγμα είναι η βελτίωση της ε, ποιότητας των υπηρεσιών Υγεία, Όχι μόνο η ε, βιωσιμότητα τους, η καλύτερη ποιότητα θα επιφέρει μεγαλό, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη παραγωγή και κατά συνέπεια μεγαλύτερη κατανάλωση. Και ε, κατά συνέπεια και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα συστήματα υγείας, αλλά και πρέπει να μιλάμε και για την ίση πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, γιατί αυτό είναι, αυτό είναι το θεμέλιο και κάτι που εμείς θεωρούμε ε, ως πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θα ήθελα να υπάρχει μέσα στην έκθεση. Η αξιοποίηση των ε, δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την μείωση της ανεργίας. Υπάρχουν τρει τομεί στου οποίου πρέπει να αναλυφθούν μέτρα. Αύξηση συζήτηση θέσεων επασχόληση στην πράσινη οικονομία, στη βάση του επίπεδου των επενδύσεων, προβλέψεις για τις ανάγκες ε, θέσεων εργασίας που βρίσκονται στη διαδικασία του πρασινίσματος και τρίτον, τον αριθμό των εργαζομένων που θα βρουν δουλειά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και από τη σκοπιά της αγοράς εργασίας θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε προγράμματα κατάρτισης που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων και προσόντων, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στους πράσινους τομείς, αλλά και στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς. Νομίζω ότι οι δυνατότητες της πράσινης οικονομίας είναι πολύ σημαντικές για την Επιτροπή μας, διότι σε κάθε συνεδρίασή μας τις αναφέρουμε και είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ε, έχουμε μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να σπαταλήσει τις δυνατότητες της αυτής και οι δυνατότητες της πράσινης οικονομίας και των πράσινων θέσεων εργασίας πρέπει να, το, να τονιστούν. Αυτή θα είναι η τομή στους θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό με τον εισηγητή και Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και θα προσπαθήσουμε να, να συνεισφέρουμε στην ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο για να υποβάλει τα δικά της σχόλια. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την DG Environment, Γιάννη Ποντέσκου. Θα ήθελα να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ενταγμένη στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για την έξυπνη ε, και βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Στην ανακοίνωση με την οποία ε, ε, η οποία αναφέρεται στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, ε, ε, στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την ανάπτυξη και αυτά δεν έχουν εξαφανιστεί. Ταυτόχρονα η ανακοίνωση δηλώνει ότι η ακόμη αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων είναι σημαντική και ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία. Δύο στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επανεπιβεβαιώνεται ε, το τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη προκειμένου να ε, σημειώσουν πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης. Αυτή η γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής ΕΝΒΗ, ε, το χαιρετίζουμε κάποιοι τρόποι για να διασφαλίσουμε ε, συγκεκριμένοι τρόποι για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Εξαμένου θα ήταν πολύ ε, χρήσιμοι. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι το 7ο σχέδιο δράσης για το περιβάλλον απαιτεί τα στοιχεία του να παρακολουθούνται στην, ε, ε, στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μας για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης. Χαιρετίζουμε τις συστάσεις της γνωμοδότησης όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη οικονομία, την, αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και αναφέρω ε, στην παράγραφο 3 της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης φυσικά η Κομισιόν ανταποκρίνεται στην έκκληση για μεγαλύτερες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ την προσοχή ε, στο επενδυτικό πακέτο που έχουμε ανακοινώσει. Υπάρχουν επενδύσεις ε, για το νερό, για την διαχείριση των, ε, των υδάτων, ε, των όμβριων υδάτων. Όλα αυτά είναι δυνατότητες. Επίσης, προβλέπεται όσον αφορά την, την πάυση χρηματοδότησης, επιδότησης των ορυκτών καυσίμων, είναι και αυτό στα σχέδιά μας. Η ετήσια έκθεση του 2015 δεν τα αναφέρει ρητός, αλλά αναφέρει την σημαντικότητα να μεταφερθεί το φορολογικό βάρος από την εργασία σε άλλους ε, τομείς που είναι λιγότερο επιβαρυντικοί για την ανάπτυξη. Και τέλος η ετήσια έκθεση τονίζει ότι προκειμένου να ενισχυθούν σε επίπεδο κρατών μελών οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει καταρτισμένο ε, εργατικό δυναμικό στους αναπτυσσόμενους ε, κλάδους της πράσινης οικονομίας. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γραμματικάκης θέλει να προσθέσει κάτι. Θα είμαι πολύ σύντομος ε, κύριε Πρόεδρε γιατί αποδείχθηκε αυτό που ζήτησα στο τέλος ότι θα είναι πολύτιμη η συμβολή, οι προτάσεις και οι ιδέες από τους συναδέλφους αλλά βέβαια και από την Επιτροπή. Πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Ε, ο κύριος Φαρία πολύ σωστά παρατήρησε για τις ευαίσθητες έτσι κατά κάποιο τρόπο επενδύσεις, για τη σημασία της κατάρτισης και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά όλα τα συμμερίζομαι ήδη, δεν τα ανέφερα στην ομιλία μου για λόγους ε, χρόνου. Και η κυρία Κονέκα είπε επίσης πολύ σημαντικά πράγματα. Λείπει, όπως είπε, η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Ε, εννοώ ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να ενισχυθούν, το λέμε αυτό στη γνωμοδότησή μας, και τα εθνικά συστήματα υγείας που είναι πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υπογραμμίζω τρεις φορές, δεν θα πρέπει να θίγονται από την οικονομική κρίση. Και βέβαια η αξιοποίηση της πράσινης οικονομίας, το τόνισε η κυρία, κυρία Κονέκα, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Ενδιαφέρον είχαν και οι παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τους ευχαρι... τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ε, κύριο συνάδελφο ή συνάδελφο ή όπως θέλετε ονομάστε τον, ε, μας διαβεβαίωσε ότι πολλά από όσα εγώ είπα στη γνωμοδότησή μου θα γίνουν πράξη ήδη γίνονται θα πω μόνο συνοπτικά ότι όπως ανέφερε πολλές φορές τη λέξη δυνατότητες η δική μας ελπίδα είναι οι δυνατότητες ε, να γίνουν πραγματικότητες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κύριε Γραμματικάκη. Τώρα μπορούμε να προσκαλέσουμε το διευθυντή της ΕΦΣΑ να πάρει τη θέση του. Ε, Οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο στη διάθεσή μας. μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 12η μεσημβρινή. 23 Φεβρουαρίου θα πρέπει να γίνει συζήτηση στην Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων. Περνάμε τώρα στην επίσκεψη του Διευθυντή της ΕΦΣΑ, Μπερνάρ Ούρλα, με τον κύριο ήρλα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της παρουσίασης του προγράμματος εργασίας Είναι διευθυντής από τον Μάρτιο του 2014, τον έχουμε ήδη συναντήσει σαν υποψήφιο. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν και θα μπορέσει να μας δώσει μια σωστή εικόνα των πεδίων παρέμβασης της ΕΦΣΑ θα μπορέσει να μας ενημερώσει για το τι κάνει η ΕΦΣΑ στην παρούσα φάση για την πρόληψη των κινδύνων των συνδεόμενων με τον ιό εμπόλα και τη σχέση μπορεί να έχουν με την τροφή. Και ταυτόχρονα θα μπορέσει να μας ενημερώσει και για τη στρατηγική της ΕΦΣΑ για την τρέχουσα περίοδο, αλλά και για ό,τι έχει γίνει στο εσωτερικό της ΕΦΣΑ, έτσι ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις ε, για την διαφάνεια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλου για τα συγκεκριμένα θέματα. και πρέπει να υπάρχει φυσικά μια πλήρης χρήση των πόρων των οικονομικών δυνατοτήτων που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σας δίνω αμέσως το λόγο για 10 λεπτά και μετά θα ξεκινήσει η συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαβία, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε μαζί σας ένα θέμα σημαντικό που είναι η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ευρώπη. Θα ήθελα καταρχάς να επιβεβαιώσω τις δηλώσει που ήδη έγινε τον Νοέμβριο, στις 10 και κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ότι η ΕΦΣΑ είναι στην υπηρεσία σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ΕΤΦΗ. Αυτό το λέει και το καταστατικό μας, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει ερωτήσεις και ε, από τους δύο ε, και τις εντολές ε, που έχει στην ΕΦΣΑ και μπορούμε και θέλω να σας διαβεβαίωσω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για καλύτερες υπηρεσίες. Έχει ένα βίο 12 ετών ο οργανισμός για να δούμε τα επιτεύγματα μέχρι τώρα να αρχίσουμε από τον ορισμό. Τι είναι η ΕΦΣΑ, πώς μπορεί να περιγραφεί. Είναι ένας επιστημονικός εταίρος για σας και για το Κοινοβούλιο για να είναι πιο ασφαλή τα τρόφιμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. 500 επιστημονικές νομοδοτήσεις εκδίδουμε ετησίως mainly ε, ε, Σε τέσσερις τομείς κάνουμε εκτιμήσεις ε, των προϊόντων και των μεθόδων και ελέγχους πριν εγκριθούν, προέγκριση. Ε, επίσης, ελέγχουμε όλη την αλυσίδα την τροφική που έχει να κάνει με την υγεία των φυτών, των ζώων, τους ρηπαντές, βιολογικούς κινδύνους, ολόκληρη την αλυσίδα της τροφής. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη στη διαχείριση ε, του κινδύνου σε περίοδους κρίσης και σε αναδιόμενους κινδύνους και επίσης ε, κάνουμε και ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να βρείτε ε, παραδείγματα πώς συνεισέφερε στο ευρωπαϊκό σύστημα ε, ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών η ΕΦΣΑ. Αν δείτε τι γίνεται με τα ζυζανιοκτώνα. Η δική μας δουλειά ήταν και οι εκτιμήσεις και η ελεγχή μας που ε, επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει κάποια χημικά στοιχεία. Επίσης, χιλιάδες ισχυρισμούς περί υγείας ελέγξαμε κατά πόσο είναι βάσιμοι επιστημονικά αυτοί οι ισχυρισμοί και μπορούν να προβάλλονται. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ε, για να ξαναγράψουμε όλη την ε, ε, ιστορία που αφορά τις προσθετικές ουσίες στα τρόφιμα. Αυτό έχει να κάνει με πολύ κέρδος στην αποτελεσματικότητα και στον εναρμονισμό των προτύπων για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι η ΕΦΣΑ συμμετείχε στην αντιμετώπιση πολλών κρίσεων, ας πούμε σε ρίχια κόλλη στη Γερμανία και στη Γαλλία ε, ή και ο ιός Μάινβερ για να σας ε, αναφέρω μερικά στοιχεία. Ε, ο ιός της υπατήτηδας α σε κατεψυγμένα σκαρπούς, κόκκινα φρούτα, βατόμουρα και ε, μπορούμε και επιγόντως να δώσουμε υψηλής ποιότητας επιστημονική συμβουλή ε, στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα. Αλλά δεν θα πρέπει ούτε να εφησυχάζουμε ούτε να επαναπαυόμαστε και να θεωρούμε ότι έτσι θα συνεχιστεί ε, και στο μέλλον η παρουσία μας όπως τα τελευταία 12 έτη. Ποιες είναι οι μελλοντικέ προκλήσεις η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, γιατί μαζί με αυτήν παγκοσμιοποιούνται και οι κίνδυνοι που συνδέονται ε, με τις τροφές και τις ζωοτροφές και όταν εισάγουμε ε, τρόφιμα, εισάγουμε και τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της ε, εξαγωγού χώρας. Άρα θα πρέπει κάθε φορά να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον και να αναθεωρούμε και τις μεθόδους που έχουμε. Επίσης, άλλη μεγάλη ε, πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή, που επηρεάζει, για παράδειγμα, τους φορείς, τους ξενιστές που μπορούν να ε, μεταφέρουν λιμώδεις νόσους ε, και μεταδόμενα νοσήματα για ζώα και για ανθρώπους για να μπορούμε στα λιμώδη νοσήματα και στα μεταδοτικά. ας πούμε, ε, ο ιός ε, ε, του καταρροϊκού πυρετού που μεταδόθηκε και στην Ευρώπη Επίσης, είναι πολύ περίπλοκος ο ρόλος της ΕΦΣΑ. Αν δείτε στα χημικά μείγματα, είναι επιστημονικές οι προκλήσεις. Δηλαδή, ε, δεν κοιτάμε μόνο τις μεμονωμένες χημικές ουσίες, ρήπαντες και ε, ζυζανιοκόνα, αλλά ε, ολόκληρες ομάδες ουσιών που ταυτόχρονα μας απειλούν γιατί υπάρχει ταυτόχρονη έκθεση. Ταυτόχρονα μειώνεται και ο πυροπολογισμός και οι πόροι που δεν μας επιτρέπουν ούτε να αυξήσουμε το προσωπικό μας ούτε τα οικονομικά μας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για την επόμενη πενταετία και πώς ε, διαμορφώνεται η προσέγγισή μας. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η ΕΦΣΑ ε, είναι να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση και μειώνονται οι πόροι. Ε, και να είμαστε έτοιμοι πάντα και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε ε, έκτακτες περιστάσεις και αναπάντεχες. Για το επόμενο διάστημα λοιπόν τρεις είναι οι βασικές για την επόμενη πενταετία στρατηγικές επιλογές. Πρώτον, συνεργασία. Θα πρέπει να είναι στον πυρήνα όλων μας των προσπαθειών. Ήδη συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με τα κράτη-μέλη σε διάφορες ε, αντίστοιχες ομόλογες οργανώσεις. Ε, όχι απλώς συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας και στα διοικητικά μας όργανα, αλλά μοιράζονται και στοιχεία τα κράτη-μέλη μαζί μας. Και θέλω να ευχαριστήσω ε, τους επιρρογνωμόνες που αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο για να εργάζονται στην ΕΦΣΑ, μαζί με την ΕΦΣΑ και για την ευρωπαϊκή υπόθεση και σας ευχαριστώ και για την πολιτική υποστήριξη της οποίας χαίρουμε στα κράτη-μέλη. Οι οργανώσεις όπου εργάζονται οι εμπειρογνώμονες τους επιτρέπουν να έρχονται οι δικοί τους εμπειρογνώμονες και να συνεργάζονται στην ΕΦΣΑ και να δίνουν επιστημονικές συμβουλές. Το μοντέλο αυτό λοιπόν με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη έχει πολλά πλεονεκτήματα, διότι έτσι μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και έχουμε και κέρδος στην αποτελεσματικότητα, δηλαδή έχουμε ένα επιμερισμό του φόρτου εργασίας και χρησιμοποιούμε τους καλύτερους κάθε φορά εμπειρογνώμονες και τους αναθέτουμε τις εργασίες. Ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στη συνεργασία, χωράει βελτίωση. Τι σημαίνει το πρόγραμμά μας, είναι μεσοπρόθεσμος στόχος αυτός, δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Και ποιος είναι αυτός. Να έχουμε ένα κοινό θεματολόγιο για την Ευρώπη, για την εκτίμηση κινδύνου. Δηλαδή, οι οργανώσεις των κρατών μελών να ξέρουν τι είναι οι προτεραιότητες, ποιες προέχουν, πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε τη δουλειά για να μην έχουμε επικαλύψεις και δίπλο δουλειές. Και ε, πρόκειται να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία. Δεύτερη στρατηγική πρωτοβουλία. Είπαμε πρώτη ήταν η συνεργασία. δεύτερη είναι η καινοτομία. Θα πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι στις επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Ε, η ΕΦΣΑ εδώ είναι πραγματικά χμή του δόρατος ε, στην επιστημονική συμβουλή, αλλά θα πρέπει να σπρώξουμε πιο πέρα τα επιστημονικά όρια και να αντιμετωπίσουμε πολύ σχηδή... Ε, προβλήματα. Σας είπα μια πρωτοβουλία που ήδη έχει ξεκινήσει πριν από λίγα χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντική για το Κοινοβούλιο και είναι ένα έργο που θέλουμε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα ε, το πρόβλημα των μελισσών, της υγείας των μελισσών που υφίστανται πολλαπλό στρες ε, από διάφορους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ίδια την επιβίωση των μελισσών. Και γι' αυτό έχουμε ένα τετραετές πρόγραμμα ένα εκατομμύριο ευρώ έχουμε εμείς επενδύσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και το εργαστήριο αναφοράς για την υγεία των μελισσών για να έχουμε μια σφαιρική καθολική προσέγγιση, να μάθουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών. Ο τρίτος τομέας που επίσης είναι σημαντικός για να προχωρήσουμε είναι η διαφάνεια, η διάβγεια. Και αυτό αφορά και αγγίζει κάτι που ανέφερε και ο πρόεδρος στην εισαγωγή του θα πρέπει η ΕΦΣΑ να μεταρρυθμιστεί και να γίνει μια ε, ανοιχτή επιστημονική οργάνωση. Τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει μόνο διαφάνεια με την κλασική έννοια, δηλαδή να μπορούν οι πολίτες και οι εταίροι μας να ξέρουν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, αλλά πάει ένα βήμα παραπέρα. Ε, διάβια σημαίνει ε, ότι συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και οι επιστήμονες που δεν συνεργάζονται μαζί μας να μπορούν να συνεισφέρουν με τη δική τους γνώση και τη δική τους πληροφόρηση στο έργο μας. Και αυτό είναι μια προσπάθεια πολυετής, έχει και κόστος. Ε, πρέπει να αλλάξουμε και συστήματα ηλεκτρονικά για να έχουμε και μια μελέτη αντικτύπου για το κόστος και το όφελος και να δούμε ποια είναι τα πιο ε, πολύτιμα στοιχεία και οι καλύτερες πρωτοβουλίες που έρχονται να προσθέσουν προς τη θεμενή αξία σε αυτό το στόχο για την διαφάνεια και τη διάφυση. Και το τελευταίο, θα πρέπει οι ε, εκτιμήσεις που κάνουμε για τον κίνδυνο να μπορούν να επαναλαμβάνονται. Δηλαδή και άλλοι επιστήμονες να είναι σε θέση να επαναλαμβάνουν και να καταλήγουν στα ίδια πορίσματα με εμάς αν θέλουν να το κάνουν Κυρίες και κύριοι, έρχομαι τώρα στο συμπέρασμα. Είναι προφανέ, πιστεύω ότι η ΕΦΣΑ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο σύστημα ασφάλεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία την επόμενη πενταετία. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους επιστήμονες, με τις ρυθμιστικές αρχές σε επίπεδο κρατών, μελών, Ευρώπης και παγκόσμιο. Ε, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις και ε, με όλους ενεχόμενους και τελικά πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να ε, δίνουμε ε, έγκυρη, αξιόπιστη επιστημονική βοήθεια. Και σε σχέση ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών εσείς και η Επιτροπή σας παίζετε σημαντικό ρόλο για την επιτυχία μας και ε, σας είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που μας δίνετε στην εκπλήρωση ε, των σημαντικών μας εντολών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά να απαντήσω σε όποια ερώτηση. Thank you to Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ξεκινάει η συζήτηση και δίνω το λόγο στον, στην ε, κυρία Πλαραγιούζο που είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας μας με την ΕΦΣΑ. Είναι χαρά που σας έχουμε ανάμεσά μας. Γνωρίζω την υπηρεσία αυτή και ξέρω περί τίνος μας μιλάτε. Υπάρχει κάτι το οποίο με εξέπληξε στην πρότασή σας. Αναφερθήκατε στο ότι αυτή τη στιγμή ε, αναφέρεστε σε ξενιστές ασθενειών. Εννοείται ε, για αναφέρεστε σε ξενιστές οι οποίοι μπορεί να μεταφέρουν ε, ασθένειες από ζώα σε ανθρώπους και αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει βέβαια είναι η τροφή και πέρα από την ευημερία των ζώων, το θέμα το οποίο εδώ είναι η διατροφική ασφάλεια και αυτή είναι η προτεραιότητά μας και η δική σας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του προσωπικού της ΕΦΣΑ ασχολείται με τα θέματα της ε, διαχείρισης είναι φυσικά οι επιστήμονες και κάποιοι έχουν αμφισβητήσει την ανεξαρτησία των συγκεκριμένων αυτών επιστημόνων. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ε, τι έχει γίνει με την περίπτωση αυτών των 15 επιστημόνων που εργάζονται στην ΕΦΣΑ. Πώς με λίγα λόγια Ε, διαμορφώνεται, συντάσσεται και πώς αποκτά αξία μια συγκεκριμένη τέτοια έκθεση. Ε, Έχουν, έχουμε ακούσει πάρα πολλές κριτικές εις βάρος της ΕΦΣΑ σε σχέση με την ανεξαρτησία των επιστημόνων, κάτι το οποίο εγώ νομίζω ότι δεν είναι, είναι αστήρικτο, δεν είναι κάτι το οποίο τεκμηριώνεται. Αλλά θα ήθελα να ελέγξω πώς ε, εσείς μπορείτε να βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά ορισμένων ε, επιστημόνων που θέλουν να ε, εργαστούν σε εσά και πώς εσείς ε, βρίσκετε τα πρόσωπα τα οποία σε μία πρώτη φάση καλούνται να αξιολογήσουν τα θέματα τα οποία εσείς εμβαθύνετε. Ε, υπάρχει μερικές φορές ε, ε, υπάρχουν εργασίες επιστημόνων οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις εργασίες τους σε σχέση με τις εργασίες τις οποίες παράγεται εσείς στην ΕΦΣΑ. Κατά τα άλλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, έχω γενικότερα θετικές εντυπώσεις. Λοιπόν, Εύη, έχετε το λόγο. Η κυρία Εύη. θα ήθελα να επαναλάβω κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες είχα καταθέσει και προηγουμένως όταν συζητούσαμε τα θέματα της απαλλαγής για τον προϋπολογισμό. και τις οποίες θα θέλω να εκθέσω εκ νέου. Ίσως και με λίγο προβοκατόρικο τρόπο. έτσι και αλλιώς τέθηκαν λίγο τα θέματα αυτά από την κυρία Γιούζο. Πώς δημιουργούνται εν πάση οι ομάδες εργασίας που φτιάχνετε και τι εγγύησει έχετε για την ανεξαρτησία των εμπλεκομένων. Είναι πραγματικά α, ανεξάρτητοι οι κριτικές οι οποίες ακούγονται από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι τεκμηριωμένες και τι είδους έρευνα κάνετε γιατί στα πλαίσια της οπτικής της μέγιστης διαφάνειας δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα θέματα των συγκρούσεων συμφερόντων που αφορούν αυτούς οι οποίοι συνιστούν τις ομάδες εργασίας. Και δεν είναι δυνατόν ε, ε, να μένουμε στη δικαιολογία ότι οι καλύτεροι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εργαστεί στις μεγάλες επιχειρήσεις κάθε φορά του τομέα. Λοιπόν, θα πρέπει ακριβώς να μην ε, ε, χρησιμοποιείται ανθρώπους οι οποίοι είχαν ή εξακολουθούν πόσο μάλλον να έχουν επαγγελματικές σχέσεις με τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Τώρα για την ανάκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην ΕΦΣΑ αυτό θα γίνει μέσω ε, διαφάνειας που θα επιτρέψει στους πολίτες και στις οργανωμένες ομάδες να εξετάζουν τις τεκμηριώσεις ε, τις οποίες δημοσιεύουν οι διάφορες ομάδες σας. Θα πρέπει να βελτιώσετε τη σχέση που έχετε με τους εκπροσώπους του κοινού συμφέροντος θα έλεγα, κάτι το οποίο ελείπει και απαιτείται να χρησιμοποιήσετε και μία πλευρά του προφίλ της, της ε, οργάνωσής σας η οποία κάνει αυτό που ονομάζουμε Open Science. Τον προηγούμενο Απρίλιο ξέρουμε ότι οθετήθηκε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να υπάρξουν ακόμα δυνατότητες ενίσχυσης της υπηρεσίας σας και να μην υπάρχουν οι σκιές του παρελθόντων. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα στα οποία συνεργάζομαι με την ΕΦΣΑ. Πολύ στενά συνεργαζόμαστε, ανάλογα με τα θέματα βεβαίω, άλλε φορέ ε, από μεγαλύτερη απόσταση. Υπάρχουν κάποια θέματα που θέλω να σα ρωτήσω. Το πρώτο είναι πολύ συγκεκριμένο για μένα και ιδιαίτερο και σα έχω ρωτήσει πολλέ φορέ. Αφορά του κανονισμού για του ισχυρισμού για την υγεία. Έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει γύρω από το είδος αυτών των ε, διαβουλεύσεων πριν από την αξιολόγηση που διατίθενταν για τις εταιρείες και ιδιαίτερα για τις ανησυχίες των καταναλωτών που, ε, που εκφράστηκαν για προϊόντα που χρησιμοποιούσαν για πάρα πολλά χρόνια που δήλθαν από μια διαδικασία ελέγχου ε, των ισχυρισμών και τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί αυτοί. Σε πολλές φορές θεωρήθηκε ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ε, ότι δεν ήταν κατορθωτό να κατανοηθεί ποιο ακριβώς ήταν ε, ο στόχος, γιατί επρόκειτο για μια νέα διαδικασία και πολλά μέλη της ε, βιομηχανίας του κλάδου της υγείας θεώρησαν ότι δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη και εσείς το δεχτήκατε αυτό, ίσως όχι με τον τρόπο που το θέτω εγώ, αλλά ε, έχετε δεχθεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε εδώ στην Επιτροπή είπατε ότι θα ήταν δυνατό και ότι θα εξετάζατε όχι να μιλήσετε με τους ετούντες άμεσα, γιατί αυτό θα ήταν υπερβολικά άμεσο στη διαδικασία, αλλά θα προσπαθούσατε να δημιουργήσετε ομάδες και να παρέχονται σε αυτές, αυτές οι συμβουλές όσον αφορά την περίοδο πριν από την έγκριση, την αδειοδότηση. Και θέλω να σας ρωτήσω πού βρίσκεστε, γιατί είναι μια εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη, σίγουρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα για τα οποία θέλω να σας ρωτήσω. Το πρώτο αφορά την απόφαση του κύριου Γιούγκερ να μην συνεχιστεί ε, η θέση του κύριου Επιστημονικού Συμβούλου, δηλαδή μια απόφαση να μην ανανεωθεί η θητεία, που νομίζω ότι είναι μάλλον αρνητική εξέλιξη. Αν εσείς ως, ε, ε ως ΕΦΣΑ θεωρήσατε ότι ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένας επιστημονικός σύμβουλος ε, και αν ε, θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σχετικά με την διαφάνεια και την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων. Είναι πάντοτε ένα θέμα που επανέρχεται σε αυτή την επιτροπή, και στην επιτροπή μας και πράγματι συζητήσαμε και για τον προϋπολογισμό και πριν από λίγο και πάλι κάποια μέλη το έθεσαν το θέμα αυτό. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω εσάς, αν είχατε την ευκαιρία αντιστοίχως να δείτε κάτι που δημοσιεύτηκε χθες την Task Force ε, για τα ζυζανιοκτώνα και τις καταγγελίες για διαφθορά ε, επιστημόνων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δια, διέρευσε για μια εκστρατεία που έγινε για, την, ε, για, να, για να αποτραπεί η απαγόρευση των ε, καρκινογόνων. Αν τελικά υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι ε, τα πράγματα είναι αμφίδρομα όσον αφορά ε, τους ε, επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Δεν είναι πάντοτε η ποσότητα των πληροφοριών αλλά και η ποιότητα. Και δεύτερον, για τα καρκινοειδή έχουμε ε, εισέλθει στην πρώτη φάση της απαγόρευσης και οι εκθέσεις από, την, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι ε, έχει μειωθεί η σοδιά κατά 30% λόγω των ζυζανίων και επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα διάθεσης των ζυζανιοκτήτων και Αναρωτιέμαι αν μπορείτε εσείς να αξιολογήσετε τις περιβαλλοντικές διαστάσεις ε, της απαγόρευσης ενός ζυζανιοκτήτου, ε, ζυζανιοκτώνου που επιφέρει την υπερβολική χρήση κάποιου άλλου. Η Κομισιόν μα είπε ότι αυτά τα δύο θέματα δεν σχετίζονται, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό, οπότε θέλω να απευθύνω σε εσά το ερώτημα. Ποια είναι, η θέση σας επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ η κυρία Πιέγκα, ο κύριος Πιέγκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε σε πολλά σημαντικά θέματα Αναφερθήκατε στο θέμα της διαφάνειας, αναφερθήκατε στο θέμα της ε, διάθεσης συνεργασίας, στην καινοτομία, αλλά σε κάτι δεν αναφερθήκατε. Και εννοώ την πρόληψη. Εγώ είμαι ιατρός και γι' αυτό η πρόληψη για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα πριν από οτιδήποτε άλλο κάθε προϊόν θα πρέπει να ελέγχεται για την ασφάλειά του για τον άνθρωπο. Ε, ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις νομοθετικές διαδικασίες γύρω από την ασφάλεια των τροφίμων. Έχουμε λάβει υπόψη μας θέματα όπως η νανοτεχνολογία ή έχουμε ασχοληθεί και με το θέμα των προϊόντων από κλωνοποιημένα ε, ζώα. Αυτά τα θέματα πώς επηρεάζουν ε, την ασφάλεια των τροφίμων. Η πρόληψη λοιπόν είναι βασικό και πάρα πολύ ε, καθοριστικό για μας θέμα. Διάβασα ένα άρθρο για μια έρευνα η οποία έγινε στην Γαλλία σχετικά ε, με την διατροφή ζώων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή μελέτη. Χρησιμοποιήθηκαν 200, ε, 200 ε, ε, ποντικοί εργαστηρίου για την συγκεκριμένη μελέτη και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Φάνηκε ότι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα σκοτώνουν πάρα πολύ απλά. Ένας μεγάλος αριθμός των ποντικών ε, έχασε τη ζωή του ε, λόγω θανατηφόρων ασθενειών κατά τη διάρκεια ε, του πειράματος. Αυτό βέβαια αφορά τους ποντικούς, αλλά θυμίζω ότι πάρα πολλά φάρμακα και πάρα πολλά καλλιντικά ελέγχονται και δοκιμάζονται σε ποντικούς εργαστηρίο. Δεν βρήκα λοιπόν απαντήσεις σε τέτοιου είδους άρθρα ερεθίσματα από πλευράς της υπηρεσίας σας. Ε, καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους άρθρα μπορεί να δημιουργήσουν και καταστάσεις πανικού ε, στα πλαίσια των αντιδράσεων. Πρόσφατα είχαμε αρκετούς θανάτους λόγω του εμπόλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις πανικού εφόσον επεκταθεί. Και αντίστοιχα κάτι μπορεί να γίνει αντίστοιχο και με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Γνωρίζω ότι τα προϊόντα, τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από γενετικά τροποποιημένη σόγια κυκλοφορούν ευρέως και γι' αυτό ακριβώς ε, έχετε μπροστά σας μια τρομακτικά μεγάλη δουλειά. Αυτά τα οποία χρειαζόμαστε δεν είναι εκ των υστέρων δράσεις, απαιτείται πρόληψη. Και αναφέρθηκα λοιπόν στα κρέατα αποκλωνοποιημένα ζώα, στην ανοτεχνολογία, και στα γενετικά τροποποιημένα γενικότερα. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Μπάρτσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θεώρησα καλό να πάρουν πρώτα το λόγο εκείνοι που ε, συνεργάζονται εδώ και χρόνια με την ΕΦΣΑ. Και αφού μίλησαν όλοι αυτοί, μπορώ να πάρω και εγώ το λόγο να μιλήσω για κάτι άλλο. Ε, πώς έχει σήμερα η κατάσταση στην ΕΦΣΑ. Είπατε κι εσείς ο ίδιος κύριε Διευθυντά ότι η εντολή σας είναι να εγγυάστε την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, για τους πολίτες στην Ευρώπη και αυτό ισχύει για όλα τα τρόφιμα. Και αφορά και τα φυτικά προϊόντα. Οπότε είναι αναντικατάστατη η ΕΦΣΑ ως οργανισμός. Έχουμε μια ερευνητική βάση και αυτή την πολύ ανοιχτή επιστημονική οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα είναι και ε, δημόσια αρχή. Και είναι ε, καθοριστικές οι γνωμοδοτήσεις σας. Ας πούμε, γενετικά τροποποιημένα φυτά ξέρουμε ότι απαγορεύονται σε κάποια κράτη-μέλη να καλλιεργούνται. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα ότι έχει ληφθεί απόφαση στο Συμβούλιο σχετικά και για σπόρους γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου. 19 χώρες εκαταψήφισαν και 5 υπερψήφισαν στο Και τώρα γίνεται λόγος για νομοθέτημα ε, σχετικό και μπορεί ενδεχομένως βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης της ΕΦΣΑ κάποια στιγμή να τα βρούμε μπροστά μας και να ε, έρθετε εσείς σε δινή θέση. ενώ μία πλειονότης και πλειοψηφία των κρατών μελών τα απορρίπτουν, μπορεί να προκύψει ε, έγκριση ε, μιας τέτοιας νομοθετικής ε, πράξης. Δηλαδή μπορεί η ΕΦΣΑ, για να το πω ξεκάθαρα, να υποχρεωθεί να υποστηρίξει τα συμφέροντα των γενετικά τροποποιημένων ε, ε, οργανισμών συγγνώμη, εις βάρος του ευρωπαϊκού συμφέροντος και των ευρωπαίων πολιτών. Το ξέρω ότι υπερβάλλω, αλλά ενδεχομένως μπορεί να έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Στο Ουγγρικό Σύνταγμα αναφέρεται ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ε, σωματική και ψυχική υγεία τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα λοιπόν δεν θα πρέπει να επιτραπούν ούτε η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων. Επιτρέπεται να γίνονται έρευνες και δίνεται γνωμοδοτήσεις ε, για πράγματα επικίνδυνα. Μπορεί να γίνει κρίσιμη η κατάσταση και μια χώρα να υποχρεωθεί να δώσει άδεια για προϊόντα, για εισαγωγές, ε, ενώ το ίδιο το Σύνταγμά της το απαγορεύει. Ή αν επικαλεστεί το, Σύνταγμά της η χώρα ε, και το τηρήσει, τότε θα της πούνε ότι παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ε, αγαθών και των εμπορευμάτων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξαφνικά οι επιστήμονες ε, θα επομιστούν μια μεγάλη σύγκρουση, θα είναι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω αν θέλουν άλλοι να λάβουν το λόγο, λέει ο ο Γενικός Διευθυντής για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Νομίζω ότι ήταν πολύ πλούσια η εισοδιά μας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομες, αλλά είναι θεμελιώδη τα ερωτήματα αυτά που θέσατε. Και ελπίζω κύριε Πρόεδρε να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να τον αφιερώσουμε στις απαντήσεις θα τις διατρέξω με, με τη σειρά που μου τέθηκαν. Ο κύριος Γιούς ρωτήσε για τις ε, μεταδιδόμενες ασθένειες, αν αυτό θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της ΕΦΣΑ ή μήπως θα έπρεπε καλύτερα να αφορά το, τον Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης ε, Νοσημάτων στη Στοκχόλμη. Εγώ μιλούσα για ασθένειες ζώων σε πρώτη φάση αν πρόκειται για μεταδιδόμενες ασθένειες και φορείς που μεταδίδουν αυτές τις ασθένειες, τότε η ΕΦΣΑ δίνει την επιστημονική συμβουλή και βοήθεια, αλλά ε, συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους από το ECDC, από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σε, σε ένα πρόγραμμα που το ε, αποκαλούμε VectorNet, ώστε να παρακολουθούμε τους, ε, τους φορείς για να ε, βελτιώσουμε την ε, ε, υγεία των ζώων και των ανθρώπων βεβαίως. Μετά ρωτήσατε για τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία και πώς λειτουργεί το, σύστημα και αυτό αφορά και άλλα ερωτήματα που έθασαν εδώ οι ευρωβουλευτές θα έλεγα, προτού ε, απαντήσω συγκεκριμένα στο ερώτημα, ότι η εγγύηση για την ε, εγκυρότητα των επιστημονικών συμβουλών της ΕΦΣΑ βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, διαχειριζόμαστε με πολύ μεγάλη προσοχή τα στοιχεία που ε, χρησιμοποιούμε στην αξιολόγηση κινδύνου. Μιλάμε για ανθρώπους, για δεδομένα επιλέγουμε δηλαδή πολύ προσεκτικά τα δεδομένα, ε, διασφαλίζουμε να έχουμε μια αποτελεσματική μεθοδολογία και επιλέγουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα μέλη αυτών των ομάδων εργασίας. Αυτή είναι, αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας. Το ποιους πόρους χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Ο δεύτερος πυλώνας που κατά τη γνώμη μου πολλές φορές ε, παραγνωρίζεται στην δημόσια συζήτηση είναι η λήψη συλλογικών αποφάσεων στα επιστημονικά πάνελ. Έχουμε 21 μέλη σε, αυτά, σε αυτές τις ομάδες επιστημονικές που θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει σαν μια μικρή επιτροπή και αυτοί οι εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη λαμβάνουν την απόφαση για την ε, επιστημονική συμβουλή της ΕΦΣΑ και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας μεμονωμένος εμπειρογνώμονας ακόμη και αν έχει κάποια κρυφή ατζέντα θα μπορούσε να επηρεάσει τους άλλους 20 προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση που είναι επιστημονικά βάσιμη. Οπότε έχουμε έναν ε, μηχανισμό ελέγχου ομοτήμων ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιστημονική γνώση ε, αξιοποιείται στην γνωμοδότηση που εκδίδουμε. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η ανοιχτότητα, ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαφάνεια. Όλα τα ερωτήματα και όλες τις απαντήσεις της ΕΦΣΑ, όλες όλα τα υλικά, τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε, τις ερωτήσεις που απαντάμε, μπορείτε να τα βρείτε στην ισοσελίδα μας. Είναι ένας από τους πιο διαφανείς οργανισμούς στην Ευρώπη, όλες οι πληροφορίες βεβαίως που ε, μας επιτρέπεται να δημοσιεύουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια ε, δεδομένα όπως τα προσωπικά δεδομένα ή τα επιχειρηματικά δεδομένα που δεν επιτρέπεται να τα δημοσιεύουμε, αλλά όλα τα δεδομένα που μπορούμε να τα διαδημοσιεύσουμε θα μπορείτε, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, για να επανέλθω στο ερώτημα του κυρίου Γιούσο, πώς επιλέγονται οι εμπειρογνώμονες. Η ΕΦΣΑ διαθέτει 10 επιστημονικά μέλη με 20 ε, επιστημονικά πάνελ με 21 μέλη και οποιοδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος μιας τέτοιας ε, επιστημονικής επιτροπής. Σε 8 ε, πάνελ βρισκόμαστε στη διαδικασία της επιλογής τους. υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει κανείς να περάσει ένα συγκεκριμένο όριο για να είναι επιλέξιμος και στη συνέχεια εξετάζουμε αυτή τη δεξαμηνή των επιλέξιμων ε, υποψηφίων όσον αφορά τις, δεξιότητες, τις δεξιότητες τους για τους, για τους βιολογικούς κινδύνους και μετά εξετάζουμε τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων για να αποκλείσουμε την περίπτωση ε, την περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων και μετά ένας κατάλογος υποψηφίων υποβάλλεται στην ε, Διευθυντική Επιτροπή του ΕΦΣΑ και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό της ΕΦΣΑ λαμβάνει την απόφαση και η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και εγγυήσεις, εγγυήσεις δεν, έχουμε, ε, δεν αξιολογούμε αυτούς τους υποψήφιους μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και προσκαλούμε παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από άλλους φορείς ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιλέγουμε τους εμπειρογνώμονες για, τα, για τις επιστημονικές μας επιτροπές. Για τις ομάδες εργασίας υπάρχει μια παρόμοια διαδικασία που εξασφαλίζει την αναξαρτησία των μελών αλλά είναι κάπως λίγο ε, πιο ευέλικτη διαδικασία γιατί μιλάμε για 5.000 ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες της εργασίας. Πώς λοιπόν διασφαλίζουμε ότι οι εμπειρογνώμονες αυτοί δεν, ε, δεν έχουν σύγκρουση συμφωνέντων. Είναι αρκετά ανεξάρτητοι. Έχουμε μια πολιτική και εφαρμοστικούς κανόνες για το πώς διαχειριζόμαστε τα συμφέροντα για να αποφύγουμε τη σύγκρουση σύμφωνων. Και αυτή η πολιτική εγκρίθηκε το 2011 από τη, Διοικη... από τη Δικούσα Επιτροπή, θα επικυρωποιηθεί και θα αναθεωρηθεί του χρόνου, θα ξεκινήσουμε δηλαδή μια αναθεώρηση του 2015, και εκεί είμαστε ανοιχτοί βεβαίως στο να συμπεριλάβουμε προτάσεις του Κοινοβουλίου, της Κοινωνίας των Πολιτών, των εμπλεκομένων, μη κυβερνητικών οργανώσεων για να αναπτύξουμε ακόμη περαιτέρω την πολιτική μας όσον αφορά την ε, ανεξαρτησία και στην πράξη οι υποψήφοι που θέλουν να δουλέψουν στην ΕΦΣΑ πρέπει να συμπληρώσουν ένα κατάλογο ερωτημάτων όπου θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα συμφέροντα που είχαν τα τελευταία πέντε χρόνια σε εννιά τομείς και στη συνέχεια ε, εμείς ενώ οι υπάλληλοι της ΕΦΣΑ αξιολογούμε αν οι εμπειρογνώμονες αυτοί είναι συμβατοί με το έργο των ομάδων εργασίας και με τον ρόλο που έχουν οι εμπειρογνώμονες σε αυτές τις ε, ομάδες. Μία αρχή είναι η εξής. Αν έχετε δουλέψει στον κλάδο ή αν έχετε παράσχει ε, συμβουλές στον ε, κλάδο, δεν μπορείτε να δουλέψετε στην ΕΦΣΑ. Αποκλείεστε. Οπότε ε, η βασική πηγή εμπειρογνωμόνων το 2012 που έχουμε στοιχεία είναι ότι 40% προέρχονται από κυβερνητικούς οργανισμούς όπως για παράδειγμα οι αρχές αξιολόγησης κινδύνου των κρατών μελών 40% προέρχονται από δημόσια ερευνητικά κέντρα 5% από πανεπιστήμια και 5% είναι ε, άνθρωποι που ε, έχουν εργαστεί, έχουν βγει στη σύνταξη και παλιότερα δούλευαν σε κυβερνητικούς ή δημόσιους οργανισμούς. Οπότε προφανώς οι υπάλληλοι του κλάδου των βιομηχανιών δεν μπορούν να δουλέψουν στην ΕΦΣΑ και αυτό είναι, ε, είναι μία από τις, από τις ασφαλιστικές μας δικλείδες. Αλλά σημαίνει και κάτι ακόμη, ότι ακόμη και αν κάποιος εμπειρογνώμονας που έχει δουλέψει ε, σε πανεπιστήμιο και έχει λάβει χρηματοδότηση από συγκεκριμένη βιομηχανία, εξετάζουμε τι είδους χρηματοδότηση ήταν αυτή και στη συνέχεια ακολουθούμε μια διαδικασία βάση κινδύνου για να αποκλείσουμε ότι αυτός ο εμπερογνώμονος θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από μια ε, σύγκρουση συμφορώντων και διατρέχει τον κίνδυνο να είναι ε, μεροληπτικός. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα πολύ όριμο και ισχυρό σύστημα που βεβαίως έχει και κόστος, πρέπει κανείς να το συντηρεί αυτό το σύστημα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κόστος που αξίζει να το αναλαμβάνουμε προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα αποτελέσματα της, ε, της ΕΦΣΑ είναι αντικειμενικά, είναι επιστημονικά βάσιμα, ότι είναι κατενοητά, ότι βασίζονται στη γνώση που υπάρχει και χρήσιμα στους ε, διαχειριστές ε, στους φορείς ε, διαχείρισης ε, κινδύνου. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό ακριβώς, να δίνουμε ε, συμβουλές σε αυτούς. Άρα τροφοδοτούμε την λήψη αποφάσεων με επιστημονικά δεδομένα. Νομίζω ότι με αυτό απάντησα και στο ερώτημα για την ανεξαρτησία, την πρόσβαση σε έγγραφα, τους ανθρώπους που εμπλέκονται ακόμα με, την, ε, με, με τους βιομηχανικούς κλάδους. Όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν στην ιστοσελίδα και κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και σε αυτή την περίπτωση η ΕΦΣΑ μπορεί να δημοσιεύσει πρόσθετα έγγραφα εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπως προσωπικά δεδομένα ή επιχειρηματικά δεδομένα τα οποία δεν μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε. Αλλά ε, να σας δώσω ένα στοιχείο. Έχουμε φέτος δημοσιεύσει ήδη 75.000 σελίδες λόγω αυτών των ετοιμάτων δημόσιας πρόσβασης ε, που έχουμε λάβει. Όσον αφορά την κυρία Γκέρλιν και του ισχυρισμού για την υγεία. Οι διαβουλεύσεις ε, πριν από την έγκριση. Νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ψηφίσει κανονισμό με βάση τον οποίο ζητείται από την ΕΦΣΑ να εφαρμόζει τα υψηλότατα δυνατά πρότυπα για, τα αποτελε... για τις αποφάσεις μας. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε τα ανώτατα επιστημονικά ε, πρότυπα που υπάρχουν Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την επικοινωνία μας με τους ετούντες για να, δούμε, για να δώσουμε πληροφορίες πώς ακριβώς θα πρέπει να υποβάλλονται τα έγγραφα. Έχουμε 8 ε, ε, έγγραφα με τα οποία εξηγούμε πώς θα πρέπει να γίνει η διαδικασία, πώς θα πρέπει να υποβληθούν τα έγγραφα, αλλά υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, έχετε δίκιο. Πρόσφατα είχαμε και μια συνάντηση με ομοσπονδίες, 15-16 ε, ομοσπονδίες για να ε, δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες. Δεν θα γίνουν κατά πρόσωπο ε, συναντήσεις μεταξύ της ΕΦΣΑ και των ετούντων. Σε αυτό δεν θα πάμε, δεν θα γίνει αυτό, αλλά Υπάρχουν ε, διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία μπορούν, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ομάδες ετούντων. Έχουν 6-7 τέτοιες συναντήσεις έχουν γίνει πέρσι. Οι ετούντες ε, μας ζήτησαν μήπως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μικρότερες συναντήσεις τις οποίες και σχεδιάζουμε και τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσουμε στην διάρκεια του 2015. Όσον αφορά τον Chief Scientific Advisor, τον ανώτατο επιστημονικό σύμβολο, η προσέγγιση της ΕΕΦΣΑ είναι ότι γενικά είναι καλό να ενισχύονται οι πολιτικές αποφάσεις με επιστημονικά δεδομένα. Και από αυτή την άποψη η κυρία Ανκλόβερ, η ε, ανώτατη επιστημονική σύμβολος, είχε ε, έναν πολύ θετικό ρόλο. Χρειάζεται ένας τέτοιος, μια τέτοια θέση, νομίζω ότι δεν είναι δικό μας θέμα, πρόκειται για πολιτικό, ε, πολιτικό ερώτημα, αλλά η Κομισιόν έχει πολλές επιστημονικές ε, πληροφορίες στη διάθεσή της, έχει τα ερευνητικά κέντρα. Υπάρχει λοιπόν αρκετό δυναμικό ε, επιστημονικό το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει η Κομισιόν. Ίσως δηλαδή και χωρίς αυτόν τον ανώτατο επιστημονικό σύμβουλο για τις ερωτήσεις σας για τη δημοσίευση τη συγκεκριμένη. Εγώ δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη όπως είπατε δημοσίευση. Είπατε ότι κυκλοφόρησε χτες αν κατάλαβα καλά. Είπατε επίσης ότι τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν αμφίδρομα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΕΦΣΑ να είναι ελεύθερη επιρροών έτσι ώστε οι ε, γνωμοδοτήσεις μας να βασίζονται σε σωστή μεθοδολογία και σε σωστές γνώσεις. Σε σχέση τώρα με όταν η ΕΦΣΑ εξετάζει ενεργές ουσίες, ιδιαίτερα για ζυζανιοκτώνα, ε, κάνουμε μια αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνεπειών και εφόσον ένα προϊόν πρέπει να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι ασφαλές για το περιβάλλον. Δεν γνωρίζω το πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκατε γιατί αν χρησιμοποιηθούν σωστά αυτά τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί έτσι ώστε να μην υπάρξουν απαράδεκτοι κίνδυνοι για το περιβάλλον. Σχετικά τώρα με την πρόληψη. Σε επίπεδο ιατρικό φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σας, η πρόληψη είναι καλύτερη. Όμως, στα πλαίσια της διαχείρισης του κινδύνου και της αξιολόγησης του κινδύνου, τα πράγματα μπορεί να λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Εμείς κάνουμε μια επιστημονική αξιολόγηση κινδύνου. Το επίπεδο του κινδύνου το οποίο δέχεται η κοινωνία είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι απόφαση της ΕΦΣΑ. Αν η αρχή της πρόληψης σημαίνει την εφαρμογή της αρχής αυτής, αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Εμείς κάνουμε αξιολογήσεις, δίνουμε δεδομένα, στοιχεία, αξιολογήσεις και προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος του κινδύνου και τα θέματα αβεβαιότητας που δημιουργούνται. Το αν θα το δεχτεί αυτό η κοινωνία είναι θέμα πολιτικό. Και νομίζω ότι είναι σωστό που στην Ευρώπη η αξιολόγηση του κινδύνου και η, και η διαχείριση του κινδύνου διαχωρίζονται. Τώρα για την μελέτη διατροφής με γενετικά τροποποιημένα από τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε με, σε μια δημοσίευση του 12 Υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις για την επιστημονικότητα αυτής της μελέτης ενεπλάκημεν στη συγκεκριμένη αυτή συζήτηση. Κάναμε μια εξαντλητική επιθεώρηση αυτής της οργάνωσης και από τα κράτη-μέλη έγιναν μελέτες και στο τέλος απεδείχθη ε, ότι ε, έπρεπε να αποσύρθει και αποσύρθηκε η δημοσίευση αυτή από το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύθηκε. Εμείς την αξιολογήσαμε και είδαμε ότι ε, υπήρχε σύμφωνη γνώμη και από άλλες υπηρεσίες εθνικού τύπου. Έρχομαι στην τελευταία σας ερώτηση για την διασφάλιση της αλυσίδας τροφοδοσίας μπορεί ε, να βοηθήσει ε, ο σωστός διαχωρισμός των ρόλων. Η ΕΦΣΑ σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα κάνει αξιολογήσεις για τις επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα βρείτε ε, στο, στις γνωμοδοτήσεις μας. Αν τώρα η κοινωνία θα τα, θα δεχτεί ή δεν τα δεχτεί αυτά τα οποία λέμε είναι άλλο θέμα. Είναι πολιτική απόφαση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αδειοδοτεί κάποια προϊόντα και να αποδέχεται κάποιους κινδύνους ή να μην αδειοδοτεί κάποια προϊόντα και να εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης λόγω οικονομικών σκέψεων, δεοντολογικών αμφιβολιών και τα λοιπά, αλλά σε επίπεδο επιστημονικό παρεμβαίνουμε και δεν προχωράμε πέρα πέρα. Το ίδιο ισχύει και για την κλωνοποίηση. Η ΕΦΣΑ έχει εκφράσει την άποψή της σε επίπεδο τροφίμικης ασφάλειας και ευημερίας των ζώων. Πέραν αυτού δεν εμπλεκόμεθα σε θέματα δεοντολογίας για το αν θα γίνει δεκτή η, η νανοτεχνολογία. Εμείς κάνουμε στην παρούσα φάση κάποιες ε, ε, επιστημονικές μελέτες. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε μεθόδους αξιολόγησης προϊόντων νανομηχανικής κτλ. Αλλά πέραν αυτού δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, για την λεπτομερή απάντησή σας. Νομίζω ότι θα σταματήσουμε πλέον εδώ. Θα πρέπει να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει μια εκδήλωση σε αυτή την αίθουσα και γι' αυτό πρέπει να μην αφήσετε τίποτα στα έδρανά σας γιατί θα απομακρυνθούν.